κρατήσετε ένα από τα τρία κουμπιά θα δούμε λειτουργεί το μηχάνημα. Η δοκιμαστική ψηφοφορία ξεκινάει. Παρακαλώ να δείτε αν δουλεύει σχεδόν ότι κανείς δεν το κάνει. Προβλέπει η διαδικασία είναι να δούμε ποιοι είναι οι παρόντες και κατά πόσο λειτουργούν τα μηχανήματα. Ωραία. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη δοκιμή και ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Συμβιβαστική. Δεν έχετε διερμηνία. Eh, Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Possiamo Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λειτουργεί. Έχετε διερμηνία. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν τη ψηφοφορία ψηφίζοντας τη συμβιβαστική 3. Υπέρ. Σηκώστε το χέρι σας παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνατε. Πάμε τώρα στην 34 υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 47 αποσύρεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τώρα στην 59 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στην συμβιβαστική 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 75 υπέρ κατά 75 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 76 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 108. Ξεκινάμε. Έλεγχος. Λείπουν δύο ψήφοι σε σχέση με τις κάρτες που εισήχθησαν. 25 κατά 27 υπέρ εγκρίνεται. Πάμε στην 109. Mauro, questo me eh. eh, se volete esporre il vostro pensiero... Αν θέλετε να εκφραστείτε, να το κάνετε αφού σας δοθεί ο λόγος και χρησιμοποιώντα το μικρόφωνο ενδεχομένω. Ορίστε, έχετε κάποια παρατήρηση. Ο κύριος Κασουλίδης, ο κύριος Ιμπίζεζικ, ορίστε. Ο κύριος Κασουλίδης. Πρόεδρε, το μηχάνημά μου δεν λειτουργεί, λέει ο πρόεδρο. Δεν λειτουργεί το μηχάνημά μου, λέει ο κ. Κασουλίδη. Θα σημειώσουμε την ψήφο σα. Μπορείτε να ψηφίσετε κόσμο στο χέρι. Ήτανε κατά η ψήφο σα. 27-26. 26 κοντράρι. 26 ψήφοι κατά. 27 υπέρ, 26 26 26 ψηφοι κατα 27 υπερ 26 κατα με μία ψήφο διαφορά περνάει. Εγκρίνεται λοιπόν η 108. Ψηφίζουμε την 111 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται μου φαίνεται η 111. Δεν είδα καλά ίσως. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 111. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 111. Chiudiamo, chiudiamo. ψηφοφορία. 20 ψήφοι κατά, 34 ψήφοι υπέρ, εγκρίνεται. Παρακαλώ σηκώντε το χέρι, διότι δεν βλέπω καλά διαφορετικά. 14 συμβαστική, τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα τη συμβαστική, 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ κατά εγκρίνεται 114 υπέρ κατά απορρίπτεται 115 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 15 υπέρ κατά εγκρίνεται πάμε στην 124 υπέρ κατά θα έλεγα ότι απορρίπτεται Ξεκινάμε λοιπόν τον ηλεκτρονικό έλεγχο για την 124. 124. Άρχεται η ψηφοφορία. 52 ψηφίσαντες, ψηφίζοντες από τους 55 που έχουμε οι κάρτες. Κλείνει η ψηφοφορία. 16 ψήφοι κατά, 38 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη, αν δεν σηκώνετε το χέρι πρέπει να μαντεύω εγώ. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Πάμε στην 128 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 129 εγκρίθηκε στη βαστική 16. Α, πάμε 132 λοιπόν. Με προφορική τροπολογία, Λούνατσεκ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 34 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά θα έλεγα Κοιτάξτε, δεν είμαι σίγουρο. Δεύτερο τμήμα τη συμβαστική 34, ηλεκτρονικό έλεγχο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, μάλλον. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν 55 του 55. Πέρα ψηφοφορία. 21 ψήφοι κατά 34 υπέρ εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική 23 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά απορρίπτεται. 197-198 υπέρ κατά εγκρίνονται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 214 υπέρ κατά θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Πάμε στη 215 υπέρ Α, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. 217. 217 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 221 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στη 224 υπέρ κατά εγκρίνεται 225 υπέρ κατά εγκρίνεται 226 υπέρ κατά εγκρίνεται 228 υπέρ κατά δεν βλέπω καλά ζητώ συγγνώμη 228 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός έλεγχος που ξεκινάει. Ψήφισαν 54 από τους 54, πέρας ψηφοφορίας, 24 ψήφι κατά 30 υπέρ εγκρίνεται. 232 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 233 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 234, όχι, καταπίπτει διότι εγκρίθηκε 233. Πάμε στη 235 με προφορική τροπολογία του κ. Σαλαφράγκα. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 237 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε συμβαστική 30 του εισηγητή σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά απορρίπτεται τρίτο τμήμα. Αν θέλετε να κάνουμε έλεγχο. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 30. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρσι οφορίε, 35 ψήφοι κατά, 19 υπέρ, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα της συμβαστική 30 υπέρ, κατά, θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Καλώς, ξεκινάμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το τρίτο τμήμα της συμβαστική 30. Ψήφισαν 52 από τις 54 κάρτες. Ωραία. Πλήρης όλοι. 29 ψήφοι υπέρ, 25 ψήφοι κατά εγκρίνεται. Τώρα πάμε, καταπίπτουν κάποιες και πάμε συμβαστική 31. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 244 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 245-246 υπέρ κατά εγκρίνεται. 247 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στη 257 υπέρ κατά απορρίπτεται. 258 υπέρ κατά απορρίπτεται 259 όχι διότι υιοθετήθηκε η συμβαστική 12 260 λοιπόν υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 33 υπέρ κατά εγκρίνεται Πάμε στην τροπολογία 266 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 267, 269, 270 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 271 προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 272 υπέρ, κατά απορρίπτεται 273 υπέρ, κατά εγκρίνεται θα έλεγα 274 υπέρ, κατά απορρίπτεται. Λοιπόν, καταπίπτουν όλες, υιοθετήθηκαν κλπ. κλπ. Α, δεν υιοθετήσαμε τη 277. Άρα πάμε στη 278 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 279 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 280. 280 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά εγκρίνεται 282 υπέρ κατά απορρίπτεται 283-284 ταυτόσιμες υπέρ κατά εγκρίνονται 285 υπέρ κατά Απορρίπτεται νομίζω η 285. Δεν είδα τα χέρια σας ξανά. 285 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. 2,85. Δεν είδα. Α, 54 ψήφισαν 26 υπέρ, 26 υπέρ, 25 κατά. Περνάει με μία. Εγκρίνεται με μια ψήφο διαφορά 285. 286 τώρα. 286 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 287 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 288 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 289 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 290 υπέρ κατά εγκρίνεται. 291, 292, 293 υπέρ κατά εγκρίνονται. 294 κατά πίπτη και 295 πάμε στην συντηρολογική σκέψη α μάλλον τροπολογία 5 υπέρ κατά απορρίπτεται 6 υπέρ κατά εγκρίνεται 7 όχι γιατί έχουν τροπολογία 6 πάμε στην 8 λοιπόν υπέρ κατά απορρίπτεται 9 υπέρ κατά απορρίπτεται 10 υπέρ κατά απορρίπτεται 11 υπέρ κατά εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται πάμε στη 15 προφορική τροπολογία του εισηγητού υπέρ κατά εγκρίνεται Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στη 17 υπέρ κατά εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά Απορρίπτεται μάλλον. Έτσι μου φαίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26 κατά διότι συμπεριλαμβάνεται συμβαστική 1. Πάμε στην τροπολογία 1, με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά εγκρίνεται και έχουμε συμβαστική 1 ίντα υπέρ Καλώς. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Αν συμφωνείτε θα ψηφίσουμε μαδικά. Θα ψηφίσουμε μαζί. Δεν συμφωνείτε. Ψηφίζουμε ξεχωριστά. Συμβαστική 1 υπέρ. Κάτα. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2, ίντα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Όλα καλύπτονται και πάμε στη συμβιβαστική, την επιστολή της Ήτρε. Λοιπόν, συμβαστική 1 της Ήτρε, ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Ήτρα 2, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τελική, άρχεται. 54 από τους 55 ψήφισαν. Ένας από τους συναδέλφους δεν δουλεύει. Λοιπόν, 52 υπέρ, μία ψήφος. Κατά συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή. Εγκρίνεται. Στρατηγική, λοιπόν. Συγχαρητήρια και στη γραμματεία που ε, Ακούσαμε τις παρεμβάσεις των συναδέλφων ότι έκανε εξοχή δουλειά γραμματεία. Επένεσαν τόσο τη δουλειά που έγινε συναδελφοί χτες. Στατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την Βαλτική θάλασσα και ο λόγος των μακροπεριοχών για το ρόλο της συνοχής. Ψηφίζουμε λοιπόν. Θα ψηφίσουμε για το συμβασμό υπερθμών 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στο 2. Υπέρ. Κατά. υπέρ, κατά, στο 3 εγκρίνεται, στο 23 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 24 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 25 με προφορική τροπολογία, υπέρ παρακαλώ, κατά, εγκρίνεται, πάλι στην προφορική τροπολογία, το 26 υπέρ, κατά, εγκρίνεται η συμβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται πάμε στην 35 υπέρ κατά εγκρίνεται 36 υπέρ κατά ε, απορρίπτεται 37 υπέρ κατά θα έλεγα εγκρίνεται 38 υπέρ κατά εγκρίνεται, 39 υπέρ, κατά εγκρίνεται, ηλεκτρονική ψηφοφορία ε, για το ψήφισμα άρχεται η ψηφοφορία. Ρε. Σκέδε 53, 52, 52. Έκλεισε λοιπόν η ψηφοφορία. Εγκρίνεται το ψήφισμα και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έκλεισαν λοιπόν οι ψηφοφορίες, πέντε λεπτά διάλειμμα πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα της μερίσιας διάταξης. Λοιπόν, συνάδελφοι, ε, ίσως να κάτσουμε σιγά σιγά. Ε, είμαστε λίγο πιο μπροστά στην ώρα, αλλά με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ε, εργαστούμε καλύτερα αν ξεκινήσουμε και νωρίτερα τη στιγμή που το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάτσετε, να ξεκινήσουν οι εργασίες μας. Ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι με αυτή τη συζήτηση ξεκινάει μια καινούργια φάση όσον αφορά την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Επιτέλους έχουμε ένα νομοθετικό κείμενο πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε. Ο ή ε, ύπατη εκπρόσωπος ε, λίγες ημέρες ε, μετά την παρουσία της εδώ για την ακρόαση τοποθετήθηκε πάνω στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και η Κομισιόν παρουσίασε κάποιες τροποποίησεις για τη χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν σήμερα καλέσαμε τον κύριο Κριστόφερσεν που εκπροσωπεί την κυρία Άστον. Καλέσαμε επίσης τον δόκτωρ Jean Jean από την ε, ε, Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και την ε, κυρία Σουκάπ από το ανθρώπινο δυναμικό που είναι αρμόδια για το καθεστώς των υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως λοιπόν γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και διότι η πρόταση είναι περίπλοκη, αλλά και πολλές φορές έχω χαρακτηρίσει την ε, πρόταση αυτή επαναστατική. Το ίδιο που έγινε και τότε με το κοινό νόμισμα. Ε, πρέπει να κάνουμε ε, μια σύγκριση του Μάστριχτ Ευρώ και της συνθήκης της Λισαβόνας εξωτερική δράση μας αναγνωρίστηκε η αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά, επειδή είμαστε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Βέβαια, τις εργασίες μας θέλουμε να τις διεξάγουμε από κοινού με την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων, Προϋπολογισμού, Ελέγχου Προϋπολογισμού και Νομικής Επιτροπής. Και γι' αυτό χαιρετίζω τους παρόντες εισηγητές, γιατί αυτές είναι επιτροπές που θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα μάλλον πριν δώσω το λόγο στους φιλοξενούμενους μας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστήσεις μας ε, προς τον εισηγητή μας, τον κύριο Μπροκ, ε, χρειάστηκε να εργαστεί αρκετές εβδομάδες, να διαβουλευθεί εργάστηκε σε στενή συνεργασία με τον ε, συνάδελφο Φερχόφστατ ε, από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και κατέληξαν σε ένα ε, πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα ήθελα λοιπόν να περάσουμε ε, στις ε, εισηγήσεις των φιλοξενουμένων μας και θα ήθελα να τους παρακαλέσω να ξεκινήσουν με πέντε λεπτά εισηγήσει για να υπάρχει κατόπιν χρόνος και χώρος για ερωτήσεις. Ε, σε εσά το λόγο, κύριε Κρίστοφερσεν. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για αυτή την ευκαιρία να πω μερικά λόγια για το σχέδιο αποφάσεως του Συμβουλίου που η Λέδη Άστον παρουσίασε μερικές μέρες αφού είχε την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις της σε αυτή την Επιτροπή. Θα ανέμενα δοθέντων των λεχθέντων επ' αυτή τη ευκαιρία ότι το περιεχόμενο της προτάσεως δεν θα αποτελούσε έκπληξη μεγάλη, διότι οι γενικές γραμμές που περιέγραψε τότε αντικατοπτρίζονται εντός της προτάσεως. Να προσθέσω επίσης ότι εν συγκρίση με τα όσα ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση του τον Οκτώβριο, στις 22 Οκτωβρίου, δεν υπάρχει διαφορά βασικά μεταξύ των απόψεων που αναφέρθηκαν τότε και των περιεχομένων τώρα στο σχέδιο αποφάσεως. Εν γέννη, να πω ότι στις 27 Οκτωβρίου στην έκθεση αυτή, μαζί με την έκθεση της Κορεπέρ που υπευλήθη στο Συμβούλιο, ότι αυτά αποτέλεσαν ακρογωνίο λίθο για την οικοδόμηση του εν λόγω οικοδομήματος. Προχώρησε ο χρόνος, κύλησε από τον Οκτώβριο. Και το Κοινοβούλιο Έτσι έχουμε κάποιες φρέσκες ιδέες παραπάνω. Κάτι το οποίο βέβαια είναι εύκολο να το αντιληφθεί κανείς γιατί όπως ε, προείπατε ο ίδιος πρόκειται για περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία. Επαναστατική. A proposal to set up a service where no blueprint. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχει μια πρόταση αναδιάρθρωσης υπηρεσίας χωρίς να υπάρχει κάποιο προσχέδιο, όπως γίνεται ας πούμε σε κάποιο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάει κανείς και λέει καλημέρα σας, αυτό θα κάνουμε. Όμως τώρα αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι κάτι πολύ παραπάνω από ότι σε μια συνήθεια υπηρεσία κάποιου Υπουργείου Εξωτερικών ε, κάποιου κράτους μέλους. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά την υπηρεσία μας αυτή, ε, θα έχουμε κάποια χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία είναι πολύ πιο ευξημένα από όσο βρίσκεται κανείς σε κάποιο Υπουργείο και θα υπάρχει επίσης επιχειρησιακή ε, δυνατότητα και όσον αφορά αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ε, θα υπάρχει επίσης κάποιο είδους ε, ιεραρχία που είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ισχύει σε κάποιο συνηθισμένο Υπουργείο από τα γνωστά. Επομένω πρόκειται για μια δομή μοναδική την οποία και εμείς τώρα καλούμεθα να σχηματίσουμε. Επίσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μας προκύψει ακριβώς η τέλεια λύση. Βεβαίως θα κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας, αλλά επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε προσαρμογές στην πορεία. Γι' αυτό και προβλέπονται μια-δυο αναθεωρήσεις, μία το 12 και μία το 14. Και γι' αυτό ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάθε φορά που θα έπρεπε να καθορίσουμε μια ακρίβεια τα διάφορα συστατικά του οργανογράμματος, γι' αυτό και δεν μπορεί να βρείτε ένα πλήρες οργανόγραμμα, μια που θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει μια κάποια ευελιξία, τόσο να έχουμε δυνατότητα προσαρμογής. Προσαρμογής στις κάθε φορά νέες εξελίξεις και για κάποια σημεία τώρα τα οποία φίξατε και ίσως είναι χρήσιμο να τα συζητήσουμε. Ε, ένα εξ αυτών είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξη, διότι πέρσι είχατε τονίσει ότι θα πρέπει να γίνει διαχωρισμό μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και των λοιπών τώρα ευθυγραμμίζεστε με την κυρία Άστον ότι δεν υπάρχει λόγος να χωριστεί ο κόσμος χωρίς ακέα και λοιπές. Οπότε και εμείς θα πρέπει να περιλάβουμε κάποια στοιχεία τέτοιας αναπτυξιακής πολιτικής καλύπτοντας στη δική μας υπηρεσία όλο τον κόσμο. Το δε βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει τώρα να επιλύσουμε θα είναι το πώς θα γίνει κάτι τέτοιο χωρίς να πέσει, Φερρυπίν. Η κάθε επιμέρους προσπάθεια. Μην πολιτικοποιηθεί υπερβαλλόντως αυτή η πολιτική ανάπτυξης. Άρα θα πρέπει έτσι να ασκήσουμε ικανοποιητικά αυτή την πολιτική. Θα πρέπει να έχουμε όλα αυτές τις μεταβλητές των αναπτυσιακών προγραμμάτων μια μεριά, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να συνεχιστεί μια αυτόνομη αναπτυσιακή πολιτική στο χαρτοφυλάκιο του αρμόδιου επίτροπου. Ο οποίος αντέσταται την προσπάθεια, αλλά φυσικά θα διατηρεί την ανεξαρτησία του. Και αυτή η πρόταση όπως είπατε για αυτόν τον κανονισμό, αυτό το σχέδιο κανονισμού είναι ε, ένας από τους βασικούς της άξονες και εν κατακλείδη θα πρέπει να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου η υψηλή εκπρόσωπο. ευθύς εξ αρχής του είπε ότι πρόκειται για ένα σύνολο, μια δέσμη μέτρων που θα πρέπει να συμφωνηθούν από όλους τους συμπλεκόμενους παρά το ότι η απόφαση προβλέπει απλώς ο γνωμοδότης του Κοινοβουλίου, γιατί γνωρίζουμε ότι η συμφωνία θα κλείσει μόνο εάν υπάρξει συμφωνία σε όλο το πακέτο. Ε, ε, ε, Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο ο κύριος Ζαν Ζαν, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα προπολογισμού. Πέντε λεπτά να έχει την καλοσύνη. Θα είμαι σύντομο, Πρόεδρε. Sur le plan, sur le plan il de tirer... Όσον αφορά τα δημοσιονομικά, τον προπολογισμό, θα πρέπει να συναγάγουμε τα... ποια είναι τα πορίσματα, τα πολιτικά. Δηλαδή, αν θα είναι μια sui υπηρεσία που θα έχει αυτονομία. Ποια είναι η συνέπεια τελικά των αποφάσεων των πολιτικών, ότι αυτή η υπηρεσία θα έχει ύπαρξη αυτόνομη όσον αφορά τον προπολογισμό, ανεξάρτητη, όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες. Αντιθέτως όμως, οι επιχειρησιακές δαπάνες, οι ειδικές δαπάνες, όπως θα διαπιστώσατε, είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό έχει κάποιες συνέπειες βεβαίω βεβαίω. Η πρώτη συνέπεια όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες είναι ότι αυτή η υπηρεσία θα είναι παρόμοια με ένα θεσμικό όργανο όσον αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό. Θα ισχύει το πρώτο άρθρο του κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί για να εμφανίζεται αυτή η υπηρεσία ούτω ώστε σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό να αποτελεί θεσμό. Δεύτερον, αυτή η υπηρεσία για τις διοικητικέ της θα υπόκειται στην απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το οικονομικό σχήμα της υπηρεσίας αντιμετωπίσαμε ένα θέμα κάπως ευαίσθητο. Ήτι. Στο βαθμό που είναι αυτόνομη αυτή η υπηρεσία και ανεξάρτητη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα δεν είναι εντός της δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επικεφαλής αντιπροσωπείων τίθεται το εξή θέμα. Σε ποιο βαθμό δίνανται να υλοποιούν ε, επιχειρησιακές δαπάνες ε, για τις οποίες δεν έχουν την άδεια διότι η, η διοίκηση Όσοι υπάρχει τώρα, η μορφή αυτή σπάει την αλυσίδα τη διοικητική. Εμεί ήμασταν δημιουργικοί, λαμβάνοντα υπόψη την ανάγκη που έχουν οι επικεφαλεί των αντιπροσωπείων πραγματικά να εκπροσωπούν απόλυτα την Ένωση στο εξωτερικό και για τις ε, επιχειρησιακές Βρήκαμε λοιπόν μια λύση. Να επανεισαγάγουμε τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών για αυτή την πτυχή των πραγμάτων, διότι αυτοί διορίζονται, όπως ξέρετε, από την ύπατη εκπρόσωπο, να επανεισαγάγουμε τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών σε μια λυσίδα διοικητική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, μέσω της οποίας αλυσίδας ως εντολών να μπορούν να συνδεθούν με την έγκριση δαπανών για για επιχειρησιακές, επιχειρησιακούς σκοπούς. Χρειάστηκε τροποποίηση ο δημοσιονομικός κανονισμός, παρουσιάσαμε τις τροπολογίες εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μερικά λόγια. Παραμένει το ισχύον σύστημα μέσω των οποίων οι γενικοί διευθυντές των υπηρεσιών των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΤΚΟ και η Γενική Διεύθυνση για τη Διεύρυνση και κάποιες άλλες γενικές διευθύνσεις περισσότερο τεχνικές ε, δίνουν τη δυνατότητα να εκτελούν οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών να χρησιμοποιούν τα κονδύλια που δίνονται στι αντιπροσωπείε. Μπορεί να δίνει σε των αντιπροσωπείων Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντολέ και οδηγίε στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Και προφανώ οι διαδικασίε εσωτερικού ελέγχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίω όλα όσα άπτονται του θέματο των οικονομικών ευθυνών, των υποχρεώσεων των επικεφαλή των αντιπροσωπείων όσον αφορά τους ελέγχους και όσον αφορά την οικονομική ε, διοργάνωση, όλα αυτά θα εφαρμόζονται. Και πιστεύω ότι η συνάδελφή μου θα παρουσιάσει ε, τα διάφορα στοιχεία σχετικά με τις συνέπειες που έχουν όλα αυτά όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής των επικεφαλής των αντιπροσωπιών. Οι κανόνες εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά αυτές τις πτυχές και μόνο αυτή την πτυχή του πραγμάτων συζητούμε εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται κυρίως οι κανόνες όσον αφορά τον έλεγχο. Ταυτόχρονα βέβαια η εξωτερική υπηρεσία θα έχει το ρόλο της τον ίδιο του ελέγχου όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες. Κατά τα λοιπά, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πολλά να προσθέσω, διότι από τη στιγμή όπου καθορίζεται σαφώ ότι οι διοικητικέ δαπάνε είναι οι δαπάνε υπηρεσίε, οι επιχειρησιακέ δαπάνε από να αποτελούν δικήμα διαχείριση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να βρεθούν λύσει τεχνική φύσεω, κάτι που κάναμε κυρίως για τι επικεφαλής των αντιπροσωπιών, για άλλα θέματα, όπως σα είπα, δευτερεύουσα σημασία, που δεν χρειάζεται να τα αναφέρω τώρα, ε, ε, παρουσίασα μια εικόνα και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο λοιπόν τώρα έχει η κυρία Σουκά, Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής ε, για Ανθρώπινους Πόρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία γενική παρατήρηση καταρχήν. Όσον αφορά τον κανονισμό προσωπικού, αυτό είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η πολιτική προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημαίνει ότι περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην απόφαση του Συμβουλίου που προβλέπει τη σύσταση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και σε μεμονωμένες αποφάσεις ε, που ε, θα λάβει η ύπατη εκπρόσωπος. Μιλάμε λοιπόν εδώ για ένα πλαίσιο Όσον αφορά τώρα το σημείο ε, κίνησης ε, για τροπολογίες υπάρχει το άρθρο 27 της ε, Συμφωνίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο αυτό βλέπουμε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης περιλαμβάνει υπαλλήλους που προέρχονται από τις υπηρεσίες του Συμβουλίου, της Κομισιόν και των κρατών μελών για να διασφαλιστεί ότι άτομα που προέρχονται από αυτές τις υπηρεσίες έχουν την ίδια ακριβώ πρόσβαση σε αυτή τη νέα υπηρεσία πρέπει να αλλάξουμε το καταστατικό διότι με βάση το ισχύον καταστατικό δίνεται προτεραιότητα ε, πρώτα ε, στους εσωτερικούς υπαλλήλου και μετά στους υπόλοιπους. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια αλλαγή και αυτή είναι και η πιο σημαντική. Ε, τώρα, στην φάση εκκίνησης, για να διευκολύνουμε την ε, ένταξη διπλωματών από κράτη-μέλη προσφέρουμε τη δυνατότητα ειδικών μέτρων που σημαίνει ότι στην περίπτωση ισοβαθμίας μπορεί να ε, προτιμηθεί ένας διπλωμάτης από κράτος μέλος γιατί επιθυμούμε ε, στην αρχή να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων. Μετά την φάση της εκκίνησης θα έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι από όλους τους θεσμούς, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αλλού και για να ε, ενσωματωθούν οι διπλωμάτες από τα κράτη-μέλη. Ε, δημιουργούμε ένα νέο προσωρινό φορέα. Εδώ εμπνευστήκαμε λιγάκι από αυτό που κάναμε για τους βοηθούς των βουλευτών. Υπάρχει λοιπόν μια ειδική κατηγορία προσωρινών υπαλλήλων και για να μπορούν οι συνθήκες εργασίες τους να μοιάζουν λιγάκι με αυτές των κανονικών υπαλλήλων, τους δίνουμε τη δυνατότητα να συνάπτουν τετραετή συμβόλαια ε, τα οποία θα μπορούν να ανανεώνονται πολλές φορές. Δεύτερον, ε, ας δούμε πώς θα διευκολύνουμε την κινητικότητα ανάμεσα στους θεσμούς. Εδώ υπάρχουν δύο σημαντικές αλλαγές. Η μία είναι ότι επιτρέπουμε τις ε, ε, μετατάξεις ανάμεσα στους διάφορους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον αυτοί συμφωνήσουν. Με βάση τον ισχύοντα κανονισμό κάτι τέτοιο αποκλείεται. Είναι λοιπόν δυνατόν να έχουμε το πηγενέλα από την Κομισιόν, το Συμβούλιο ε, και την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, μετά από συμφωνία μεταξύ τους. Βεβαίως αυτό θα είναι κατά εξαίρεση περίπτωση και θα δούμε μετά πώς θα το ρυθμίσουμε. Και κάτι άλλο πάλι για να διευκολύνουμε την κινητικότητα. Είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε δικαίωμα επιστροφής. Δηλαδή όλοι όσοι θα είναι στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, θα μπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους θέση και θα έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα όπως και οι εσωτερική υποψήφοι. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ειδική περίπτωση του προσωπικού που εργάζεται στις ε, αντιπροσωπίες. Ξεκινάω με τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών. Όπως είπε και ο συνάδελφός μου, κύριο Ζαν Ζαν, Συμφωνήθηκε λοιπόν ότι ο διορισμός των επικεφαλής αντιπροσωπιών θα γίνει βεβαίως από την ύπατη εκπρόσωπο, αλλά με βάση ε, έναν κατάλογο επιλογής, ένα short list, ε, με τον οποίο κατάλογο θα πρέπει να συμφωνήσει και η Κομισιόν. Όσον αφορά τώρα το προσωπικό της ε, Κομισιόν που θα εργάζονται στις αντιπροσωπείς, θα τους επιτρέψουμε να λαμβάνουν εντολές από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας και παράλληλα προβλέπουμε για τα ε, καθήκοντα της Κομισιόν που ε, θα πρέπει να αναλαμβάνει επικεφαλής αντιπροσωπείας, εκεί θα μπορούν να λαμβάνουν εντολές και από την Κομισιόν. Αν θέλετε λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που έχουμε στον κανονισμό προσωπικού. Όσον αφορά τη διαδικασία, θέλω να σας πω ότι προς το παρόν δεν έχουμε καταθέσει μια πρόταση, γιατί διαπραγματευόμεθα με τα συνδικάτα. Ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις την προηγούμενη εβδομάδα και μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα, θα πρέπει να διαβουλευτούμε με την Επιτροπή Προσωπικού και μόνο μετά η Κομισιόν θα μπορεί ε, να ε, υιοθετήσει την τυπική της πρόταση, η οποία βεβαίως θα διαβιβεστεί στο Συμβούλιο και ε, στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε την κυρία Σούκα και ξεκινάμε με τον κύριο Μπρόκ. Ε, ίσως μπορείτε να περιοριστεί σε δύο λεπτά. Καλό θα ήταν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ε, όλο αυτό το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχει μόνο συμφωνία ανάμεσα ε, στην Κομισιόν, το Συνοβούλιο και το Κοινοβούλιο όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα άσκησης βέτο. Ε, το που έχει σημασία είναι να υπάρχει μια κοινή βάση εμπιστοσύνη. Κατά την άποψη του Κοινοβουλίου υπάρχουν δύο θέματα που πρέπει να επιτευχθούν. Πρώτον, συμφωνία με όλου για να υπάρχει μια εύρυθμα λειτουργούσα ε, ε, έκφρασή μας και αντιπροσωπεία μας προς τα έξω. Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Το δεύτερο είναι τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον προπολογισμό, στον έλεγχο, στην απαλλαγή, αλλά και τα πολιτικά δικαιώματα, ε, τα δικαιώματα λήψη αποφάσεων ε, που προβλέπονται. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει μια σειρά προβλημάτων ε, και εδώ θα ήθελα λιγάκι να μου διευκρινίσετε ε, πριν ακριβώ πρόκειται, γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει ακόμα να διαπραγματευτούμε. Review clause 2012-2014, ε, καλή ιδέα αυτή, όμως το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να λυθεί τώρα το πρόβλημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σημαντικά θέματα δεν θα δεχθεί να παραγωνίζεται λόγω της ρήτρα αναθεώρησης review clause. Και εδώ μια ερώτηση προς τον κύριο Μπλανσόν. Ε, και η κυρία ε, Κρέσλε νομίζω θα ρωτήσει και αυτή. Μήπως μπορείτε να μας ε, εξηγήσετε πώς η τροποποίηση του άρθρου 1 του Δημοσιονομικού Κανονισμού τα δικαιώματα ελέγχου και προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υφίστανται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο αν η υπηρεσία αυτή να ανήκει στην Κομισιόν γιατί για μας ε, είναι πάρα πολύ απλό και αυτή είναι και η θέση μας. Αν είναι ε, μέρος της Κομισιόν ή αν ε, έχει ένα καθεστώς όπως η Όλαφ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, αν θέλετε άλλη λύση, θα πρέπει να μας ε, πείσετε πώς θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επ' αυτού πρέπει να σας πω ότι δεν έχω ακόμα επαρκείς διαβεβαιώσεις. Ένα άλλο θέμα ε, θα ήθελα να το ε, απευθύνω κυρίως τον Χριστόφερσεν, δηλαδή με ποιον ακριβώς τρόπο διασφαλίζονται τα πολιτικά δικαιώματα του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν πρόκειται για αποστολές, εντολές, διαπραγματεύσεις, θέματα που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση στρατηγικών, με την κατάρτιση της εξωτερικής πολιτικής, με ποιον ή ακόμα αν θέλετε και το θέμα των διορισμών Πώ ε, Πώς ακριβώς θα ε, συμπεριλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ποιο επίπεδο θα γίνεται αυτό ε, για να περάσουμε και στην ε, πρακτική συνεργασία. Γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αναφέρεται ούτε στον κανονισμό προσωπικού, ούτε στον ε, δημοσιονομικό κανονισμό, ούτε στον κανονισμό του Συμβουλίου. Για μας αυτό είναι ένα ερώτημα κλειδί, όπως επίσης και το θέμα του προϋπολογισμού και από τι μάλλον από εκεί θα συναρτάται η δράση μας κατά το μέλλον. Τέλος, για τον κανονισμό του προσωπικού, staff regulation. στο συνθήκη δεν αναφέρεται ότι ένας από τους ε, τρεις ε, φορείς ε, θα πρέπει ο κάθε ένας από αυτούς και τα κράτη-μέλη να διαθέτουν το ένα τρίτο. Όχι, αυτό δεν αναφέρεται στη συνθήκη. Λέει μόνο τρεις πηγές, από εκεί θα προέρχονται πάλι, υπάλληλοι, χωρίς να διευκρινθεί τίποτα. Και αυτό δεν ξέρω, είναι ένα τρίτο κομισιόν και ένα τρίτο ε, συμβούλιο γιατί ε, όπως είπε και ο κύριος ε, Αλμέιντα αλλά και ο κύριος Κριστόφερσον είπαν ότι αυτά δεν είναι απαραίτητα θέματα της ΚΕΠΑ αλλά είναι άλλα θέματα που έχουν σχέση με την κοινοτική πολιτική. Μήπως λοιπόν οι κοινοτικοί υπάλληλοι από την Κομισιόν τελικά καταλήξουν να είναι στην μειοψηφία και να επικρατήσουν άλλες πλειοψηφίες. Θα ήθελα μια διευκρίνηση επ' αυτού και μια διευκρίνηση όχι μόνο για τους ε, ε, συμβασιούχους από τα κράτη-μέλη, όχι μόνο για τα κριτήρια που θα ισχύσουν ως προς την επιλογή τους. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι καλό να ακολουθηθεί ε, ως πρότυπο το καθεστώς και των βοηθών των ε, Ευρωβουλευτών. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω ότι οι Ευρωβουλευτές σίγουρα ε, θα απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το παλιό καθεστώς των βοηθών. Γι' αυτό σας λέω και εγώ καλύτερα να δείτε λιγάκι την πρακτική, το τι ισχύει. Είπατε ότι αν κρυθεί απαραίτητο μπορούν να ανανεωθούν οι συμβάσεις. Ποιος το αποφασίζει, το κράτος μέλος ή είναι η απόφαση του υπαλλήλου. Αν αποφασίζει το κράτος μέλος, τότε μήπως η αφοσίωση προς την πατρίδα είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι η αφοσίωση προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και αν μιλάμε για το 1 τρίτο, των υπαλλήλων, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει αυτό που θα λέγαμε αφοσίωση στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, τουλάχιστον από το 1 τρίτο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπροκ και το... Συγγήτρια την Επιτροπή Προπολογισμού, η κυρία Γκρέστα έχει το λόγο. Τρία-τέσσερα λεπτά ενδεχομένω έχετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ζων Ζων μίλησε για την ε, ε, πραγματικότητα. Εγώ θέλω να πω ότι Υπάρχουν ε, προτάσεις ε, που έχουν κατεθεί διότι στις ε, προτάσεις βλέπουμε ότι επικρατεί το ευρωπαϊκό ε, δημοσιονομικό δίκαιο. Αυτό όμως που ισχύει τώρα προέκυψε μετά από σκάνδαλα και γι' αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάποιες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου ε, προϋπολογισμού υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται για να συσταθεί μια υπηρεσία εκτός της Κομισιόν. Όλα αυτά τα ε, προβλήματα και οι περίεργες κινήσεις θα ήταν περιτά αν, ε, όπως σας είπα, είχαμε ξεκινήσει διαφορετικά. Ο ύπατος εκπρόσωπος είναι εκείνο που δίνει τις εντολές και δαπανά τα χρήματα της ε, Κομισιόν. Ε, για μας αυτό δεν είναι γνωστό. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι με κάτι τέτοιο. Ε, εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι οποτεδήποτε υπάρχει ανάμειξη αρμοδιοτήτων, αυτό δεν είναι καλή ιδέα, γιατί τελικά λείπει ε, η τελική ευθύνη, ο ένας και μόνος υπόλογος. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι αυτά τα πράγματα ε, πρέπει να δοκιμαστούν καταρχήν. Και θεωρώ ότι αγνοήθηκαν κάποια στοιχεία του προπολογισμού από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα. Ε, στο νέο αυτό δίκαιο έχουμε conflict of priorities, κάτι που αναφέρεται καινούριο, σύγκρουση προτεραιοτήτων. Αυτό δεν το γνωρίζαμε. Τι είναι αυτό. Ε, γι' αυτό φταίνε όμως η πολιτική. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με την δημιουργία ε, μιας παράλληλης οργάνωσης ε, που αν ήδη τώρα κρίνεται ανεπαρκής καταλαβαίνετε τι θα πιστέψει ο φορολογούμενος. Έχουμε τη λύση ότι αρμόδια για να δίνει εντολέ είναι η ύπατη εκπρόσωπο. Μέχρι τώρα κανένα επίτροπο δεν είχε δυνατότητα να δίνει εντολέ. Και αυτό δεν είναι καλό ούτε για την κυρία αυτή, την ύπατη εκπρόσωπο, η οποία τελικά φέρει ευθύνη τεράστια για πράγματα που ούτε καν μπορεί να γνωρίζει. Μετά, στην απαλλαγή. Αυτή τη στιγμή, με βάση συνθήκη, η Κομισιόν μόνο απαλλάσσεται από εμά. Για όλου τους άλλου θεσμού έχουμε προβλέψει την πολιτική απαλλαγή και κατ' ουσίαν θέλαμε να αποφύγουμε να ορίσουμε τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Αλλά κατ' ουσίαν δεν υπάρχει απαλλαγή κανό άλλου οργανισμού πλην τη Κομισιόν ε, εμείς ε, ως Κοινοβούλιο δεν χρειαζόμαστε καμία άλλη διαβεβαίωση πέρα από αυτά που αναφέρονται. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να ε, προσέχουμε ιδιαίτερα τα θέματα της ε, έρευνας και της ανάπτυξης. Στην Κομισιόν υπάρχει μία ιεράρχηση Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα όπου η Κομισιόν μπορεί να δαπανίσει χρήματα. Το ένα είναι Country Allocations, το άλλο είναι Continental and Regional Strategic Papers και το τρίτο είναι Nips and Pips και το τέταρτο είναι Activity Program. Και στην πρόταση της κυρίας Άστον αναφέρεται ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης φέρει ευθύνη για τρεις από τέσσερις αυτούς τομείς, άρα δηλαδή η Κομισιόν τελικά είναι μόνο το εκτελεστικό όργανο. Για μας όμως εδώ πρόκειται για δις ευρώ. Άρα ε, και αυτό ε, πρέπει κάπως να το εφαρμόσουμε στην ε, πρακτική. Και γι' αυτό λοιπόν δεν θα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι μέχρι τώρα είχαμε τον έλεγχο και την απαλλαγή της Κομισιόν. Το θέμα τώρα του προσωπικού. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δαπανάνε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Τώρα αν στο μέλλον έχουμε τους διπλωμάτες που δαπανούν χρήμα των Ευρωπαίων φορολογούμενων, εκεί τι θα γίνει. Αν γίνει κάποια τασταλία, πώς θα ακριβώς θα ρυθμιστεί αυτή γιατί ε, τις ε, λύσεις αυτές ε, δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε στους διπλωμάτες, δεν έχουμε πρόσβαση αυτούς και ας πούμε ένας Γερμανός υπάλληλος ο οποίος είναι για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης στη Νότια Κορέα και αυτός παραβιάσει το δίκαιο περί δημοσιονομικών υπερπιπλογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα τον δικάσουμε, πού ευθύνεται και με ποιο δίκαιο. Κατόπιν, θέματα που αφορούν στον προϋπολογισμό ε, και την κυρία Άστον. Εγώ πιστεύω ότι για μας ε, θα ήταν σκόπιμο ε, προτάσεις που έχετε καταθέσει να αποσυρθούν εφόσον είναι τόσο λεπτομερείς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό. Ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε επί της αρχής και να μην υπάρχουν τόσες πολλές λεπτομέρειες γιατί μετά όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή ε, δεν θα μπορούμε να εφαρμόσουμε ορισμένα θέματα. Αυτά είχα να πω από αυτού και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ο Γκουαλτίαρη, εκπρόσωπος Επιτροπής Πολυπολογισμών. Για τεσσερα λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα έλεγα ότι τώρα, αφού προερχόμαστε από μια συζήτηση στο Επιτροπή Προπολογισμών του θέματο, η πρόταση, το πακέτο, ενδέσμη προτάσεων ε, έχουν σαφή βάση. Ε, προσπαθούν να συγκεραστούν δύο απαιτήσει. Δηλαδή, από τη μία η απόφαση η υπηρεσία αυτή να βγει εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η άλλη απέτηση διαφύλαξης των προνομίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό γίνεται μέσω περίπλοκου μηχανισμού που διαχωρίζει τις διοικητικές δαπάνες που είναι εκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι λειτουργικές εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι επικεφές των αντιπροσωπιών έχουν διπλή ιδιότητα κατά κάποιο τρόπο. Είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας αλλά είναι και υπεύθυνοι εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, ε, εκτέλεση του προπολογισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως ότι αυτή η πρόταση, αυτό, αυτή η ευρυδική λύση δημιουργεί προβλήματα. Εγώ διαφωνώ με την κυρία Γκλέσλε. Δεν βλέπω αυτά τα προβλήματα τόσο πολύ όσον αφορά το δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον αφορά προπολογισμό. Αντίθετα, θα έλεγα ότι ως διαφάνηκε από την προηγηθή σα συζήτηση ότι υπήρχε ένα τμήμα αυτόνομο, ξεχωριστό, διοικητικό της υπηρεσίας και αυτό καθιστά πιο διαφανή, πιο σαφή την διαδικασία της απαλλαγή. Όμως υπάρχουν και προβλήματα αποτελεσματικότητα, θα έλεγα. Οπότε είναι κατανοητό το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μιας επιτροπής, μιας υπηρεσίας που να επισέχεται ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας όχι μόνο ένα πρόβλημα διοικητικής φύσεως, συνοχής και διοικητικής αποτεσματικότητας και συνοχής μπροστά μας, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ιστορικοπολιτικό, που δεν είναι μόνο το πρόβλημα της συνένεσης που ήδη έδωσε η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την θέληση ε, του Συμβουλίου να η Επιτροπή αυτή, η υπηρεσία να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ιστορικό πολιτικό πρόβλημα που ε, προέρχεται από τη νέα διάσταση της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ε, της κοινή ασφαλείας, και της, ΚΕΠΑ και της ΚΕΠΑ δηλαδή. Είναι μια διάσταση που είναι δύσκολο να, να κοινωτικοποιηθεί άμεσα. Άρα είναι ένα πολιτικό πρόβλημα που έχει μπροστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, να καταλάβουμε αν αυτό το υβριδικό μόρφωμα θα πρέπει να τίνει προς επανεθνικοποίηση του κοινοτικού ή ένα ευρύδιο που θεωρούμε σαν ένα στάδιο προσταδιακής κοινοτικοποίησεως της εξωτερικής δράσης ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ενώσης. Αν το Κοινοβούλιο τοποθετείται προς αυτή την κατεύθυνση και οι διαπραγματεύσεις βασίζονται επ' αυτού, πιστεύω ότι θα πρέπει αμέσως να εντοπιστούν κάποια προβλήματα συγκεκριμένα που τίθενται. Το πρώτο πρόβλημα είναι του ελέγχου περισσότερο, του πολιτικού ελέγχου από ότι του προπολογισμού πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν κενά από αυτή την έποψη, όχι μόνο στην πρόταση, αλλά και στο συνολικό πακέτο προτάσεων. Θα έλεγα πάνω απ' όλο ότι θεωρώ πραγματικά ανησυχητικό και πολύ δυσνόητο το ότι προτείνεται διάλογος με το Κοινοβούλιο και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία ανανέωση της διαθεσμικής συμφωνίας επί του προπολογισμού που όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του προπολογισμού της ΚΕΠΑ προτείνει ακριβώς το παλιό σχήμα πριν τη Λισαβόνα και αυτό πραγματικά είναι απαράδεκτο. Και μετά υπάρχουν και άλλα θεμελιώδη σημεία. Ένα θεμελιώδε θέμα είναι πολύ δύσκολο να συζητείτε μία πρόταση από την οποία λείπει το παράρτημα. Διότι αυτό το θέμα του ποια τμήματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταφέρονται στην υπηρεσία είναι θεμελιώδη σημασία που αφορά και το ρόλο, την αυτονομία των αναπτυσιακών πολιτικών. Διότι από αυτή την έποψη πραγματικά λυθεύει ότι το σύστημα Joint Key που αναφέρεται εγγυάται ότι η υπηρεσία διαχειρίζεται τον προγραμματισμό των προγραμμάτων των αναπτυξιακών για λογαριασμό του επιτρόπου που έχει την, το ρόλο λήψης πολιτικών αποφάσεων. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνοι που θα υλοποιούν αυτό το έργο, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά, είναι αυτοί που κάνουν στην DG, Relex και ΤΕΒΕ e τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα υπάρχει διάχυση αυτή τη κληρονομιά τη επαγγελματική και των αρμοδιοτήτων και αυτονομία όσον αφορά την ανάπτυξη. Και υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά προβλήματα που ήδη αναφέρθηκαν από τον συνάδελφο Μπροκ, επί των οποίων θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση στεναρή. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη, θα δώσω το λόγο ακολουθώντας τη σειρά που έδωσα στην αρχή της ε, συνεδριάσεως. Λοιπόν, ανάλογα με τις αρμοδιότητες σας, μοιραστείτε τις απαντήσεις, αλλά ο καθένας παρακαλώ 3-4 λεπτά το πολύ για τις απαντήσεις που θα δώσετε. Ο κ. Κριστόφερσεν έχει το λόγο πρώτος. Thank you very much. Um, I will start with, um... Σας ευχαριστώ. Για να αρχίσω με αυτό το οποίο ερώτησε ο κύριος ε, Μπροκ για την ε, πολιτική ευθύνη και υποχρέωση σε λογοδοσία. Βεβαίω και θα πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδους ε, υποχρέωση στην διαδικασία και στη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε, γι' αυτό είναι βασικό πολιτικό συστατικό. Η Πάτη Πρόσωπος ξεκάθαρα τόνισε ότι η υπηρεσία η οποία τώρα υπάρχει θα προσαρμοστεί στην καινούργια. Και απάντησε με σαφή τρόπο σε σχέση με κάποιους ε, διορισμούς υψηλών υπαλλήλων σε σχέση με την συνεργασία και έγκριση εκ μέρους του Κοινοβουλίου, είδαμε και σήμερα το πρωί τι έγινε. Και η διαδικασία αυτή θα ισχύσει και για κάποιες υψηλέ, άλλες θέσεις ε, διπλωματών ψηλού βαθμού. Επίσης, ξέρει πολύ καλά ότι το Κοινοβούλιο είναι η αρμοδία για τον προπολογισμό αρχή και ότι επομένω θα χρειαστούν κάποιες κινήσεις επίγουσε ούτω ώστε το κοινοβούλιο να μπορέσει να συμπλέψει. Είναι αυτά τα στοιχεία επομένω, τα οποία θα διαβούν τη λειτουργία της νέας εξωτερικής υπηρεσίας. Βέβαια το θέμα είναι ότι έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με το τι γίνεται αλλού σε άλλους χώρους. Δηλαδή υπάρχει ζήτηση για παροχή συμβουλών όσον αφορά τις διεθνείς ε, συμβάσεις. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κάποιε αποφάσεις επίσης επιτροπολογίας για κάποια αναπτυξιακά προγράμματα που ε, επίσης απαιτούν ε, παροχή συμβουλών και είπε από αυτόν ο κύριος Άστον ότι ο σωστός χώρος για τέτοιες συζητήσεις είναι αυτό, αυτό το καινούργιο όργανο των παράλληλων συζητήσεων που σαν πλαίσιο θα αρχίσει σύντομα να λειτουργεί. Για αυτό το M3, το 2 τρίτα, δεν κατάλαβα πολύ καλά, γιατί μια φορά και έναν καιρό, τότε που είχε την Προεδρία η Σλοβενία, λέγεται ότι το N τρίτον του προσωπικού θα προέρχεται από την γραμματεία του Συμβουλίου κατά το οποίο καταργήθηκε, το 1 τρίτον είπαμε από τα κράτη-μέλη και το 1 τρίτον υπαλλήλου τη Κομισιόν. Επομένω, τουλάχιστον 1 τρίτον θα είναι από τα κράτη-μέλη και αν δείτε τα στοιχεία προκύπτει σαφώ ότι η πλειοψηφία του προσωπικού προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασικά από εκεί θα γίνει η προσλήψη. Και Στη βάση του σημερινού προσωπικού, αν κάνουμε κάποιου χοντρικού υπολογισμού, πάμε στον αριθμό των 600 700 υπαλλήλων τη Κομισιόν που θα πάνε στην υπηρεσία αυτή εξ εξαρχία. 55 από την γραμματεία του Συμβουλίου και κάποιοι από την υπηρεσία ασφάλειας και άλλους 200 από το στρατιωτικό προσωπικό. Εν πάση περιπτώσει, η προεχόμενη την Κομισιόν θα είναι στο 50% τουλάχιστον. Άρα δεν έχουμε εκεί πέρα κάποια αμφιβολία για το τι θα γίνει και επίση τι θα γίνει με την ε, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Καταρχήν, οι διευθύνσει, τα τμήματα, τα γεωγραφικά θα έρθουν στη δική μας υπηρεσία από την διεύθυνση. Σαν ανάπτυξη δεν θα πάνε ούτε στην ΡΕΛΕΞ, ούτε στην γραμματεία του Συμβουλίου. Αυτοί ας πούμε που ασχολούνται με την ε, Αφρική θα έρθουν σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρίστοφερσεν για τρία-τέσσερα λεπτά. Το λόγο έχει ο κύριος Ζαν Ζιάν. Euh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα επιμείνω. Στο εξής. Όσον αφορά τις επιχειρησιακές δαπάνες. δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά το ρόλο της Επιτροπής. Και αυτό δυνάμει των όσων προβλέπουν οι συνθήκες σε αυτό είναι ξεκαθαρές. Συγκεκριμένα τώρα το 317, εκεί όπου ορίζεται ότι η εκτέλεση του προπολογισμού γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο ότι ο δημοσιονομικό κανονισμό προβλέπει συγκεκριμένη αρμοδιότητα σε περίπτωση που κάθε θεσμικό όργανο ε, μετέχει στην εκτέλεση προπολισμού για τι ίδιε δαπάνε, δηλαδή τι διοικητικέ. Άρα, πρώτον, όσον αφορά τι λειτουργικέ επιχειρησιακέ δαπάνε, όσον αφορά τον έλεγχο και όσον αφορά την διαδικασία της απαλλαγής όλα όσα σήμερα ισχύουν θα συνεχίσουν να ισχύουν και αύριο. Επομένως, το Κοινοβούλιο δεν θα αλλάξει τίποτα ρόλο του σε σχέση με ασχήνουν σήμερα, τώρα όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες. Η κυρία Κρέσλα έχει δίκιο, όπως και ο κύριος Μπροκ. Αυτό ορίζει η συνθήκη. Ότι Σύμφωνα με το άρθρο 119 το Κοινοβούλιο παρέχει την απαλλαγή στην Κομισιόν. Όμως θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι στην πράξη το Κοινοβούλιο παρέχει χωριστά την ε, απαλλαγή σε κάθε θεσμικό όργανο. Κύριε Γκρίσλε θεώρησε ότι είναι πολιτική η απαλλαγή. Και ο Δημοσιονομικός Γενικό προβλέπει ότι τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να τηρούν κατά λεπτό τις διατάξεις της απαλλαγής. η οποία σε κάθε θεσμικό όργανο παρέχεται χωριστά και σας θυμίζω ότι η κυρία Άστον μίλησε στο κοινοβούλιο ξεκάθαρα δεν άφησε κανένα σημείο αδιευκρίνιστο σε σχέση δηλαδή με το ότι θα επαχθούμε και ως εξωτερική υπηρεσία στην διδασκαλία της απαλλαγής όσον αφορά τις ε, πιστώσεις που θα πρέπει να διαχειριστούμε. Άρα γι' αυτό νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Και αυτό είναι το βασικό θέμα, Πρόεδρε. Τώρα τι άλλο αναφέρθηκε. Α, η κυρία Γκρέσλε μα είπε κάτι για τον προγραμματισμό, για την διαχείριση των χρημάτων, γιατί για άλλη μια φορά, εν προκειμένου, πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ του προγραμματισμού καθεαυτού αυτού και από την άλλη μεριά τη διαχείριση των ε, λειτουργικών εξόδων. Αυτά τα οκτώ δίσκοπη κυρία Γκρέσλε, που θα συνεχίσουν να τα διαχειρίζονται οι της Κομισιόν με την ισχύουσα διαδικασία δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτό είναι σαφώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, το λόγο έχει η κυρία Σούκα, Σούκα, Σούκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να διευκρινίσω κάτι πράγματα, μερικά πράγματα. Το 1 τρίτα, 2 τρίτα, αυτό δεν αναφέρεται πουθενά ε, στον κανονισμό προσωπικού. Αυτό ε, αντιμετωπίζεται ξεχωριστά εκτός ε, κανονισμού προσωπικού. Κοιτάξτε, εγώ έκανα μία σύγκριση λιγάκι με τους βοηθούς των βουλευτών, αλλά πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτό αφορά μόνο τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Δηλαδή, για τους εθνικούς διπλωμάτες χρησιμοποιούμε μια ειδική κατηγορία προσωρινών υπαλλήλων υπαλλήλων και οτιδήποτε έχει σχέση με την εξωτερική υπηρεσία, αυτό εξετάζεται τελείως ξεχωριστά. Δηλαδή εκεί σταματάει η συγκρισιμότητα. Είναι μόνο το θέμα της μεθόδου και τίποτα άλλο και σας διαβεβαιώ επ' αυτού. Όσον αφορά τώρα την παράταση, την ανανέωση των συμβολέων. Ποιος αποφασίζει η ανανέωση των συμβολέων, αποφασίζεται από την ύπατη εκπρόσωπο, αλλά η προϋπόθεση είναι ε, το κράτος μέλος ε, να ε, δώσει τη συγκατάθεσή του. Άρα δηλαδή κοινή στάση απέναντι στην ανάμεσα στο κράτος μέλος και στην υπατή εκπρόσωπο. Κυρία Κρέσλε, αναφέρθηκε στο ότι οι ε, κοινοτικοί διπλωμάτες ε, θα χρησιμοποιούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό ε, στον προσωρινό κανονισμό και προβλέπουμε ότι αν τελικά η ε, αρχή, η διορίζουσα αρχή απαιτήσει πειθαρχικά μέτρα, τότε αυτά τα μέτρα θα πρέπει να δρομολογηθούν από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Νομίζουμε λοιπόν ότι είμαστε καλυμμένοι. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σούκα και πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων και θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο ε, για δύο λεπτά στον κύριο Θα Δίνουμε το λόγο πρώτα στους σκιώδη ηγητές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω λιγάκι σε κάτι ε, το οποίο το θεωρώ μια σουρεαλιστική κατάσταση. Η συνάδελφος κυρία Γκρέσλε είναι εμπειρογνώμων για θέματα προβλησμού, όλοι την εκτιμούν και λέει εδώ ότι παραβιάζεται κατάφορα το δίκαιο του προπολογισμού, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο θα λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία. Η Κομισιόν μας λέει ότι δεν αλλάζει τίποτα, η Κομισιόν έχει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την εφαρμογή και τον έλεγχο του προπολογισμού. Δεν είναι ότι είμαστε δύσπιστοι, μόνο που εδώ ε, έχουμε ένα σουρεαλιστικό διάλογο. Ε, καθαρά πολιτικά είπατε εκπρόσωπο και το είπατε κι εσείς, είπε λοιπόν με σαφήνεια ότι υπάγεται στην απαλλαγή. Το θέμα είναι νομικά πώ θα γίνει αυτό και ισχύει αυτό που λέει η κυρία Κρέσλε ότι υπάρχει πράγματι παραβίαση του δικαίου περί προπολογισμού και αν ναι θα πρέπει να βρούμε έναν δρόμο για να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια ότι εδώ έχουμε μία σαφή πολιτική δέσμευση. Ο κύριο Μπρόκ είναι το πρώτο ε, που είπε, ρώτησε την κυρία Άστον, εξακολουθεί να υπάρχει απαλλαγή, θα εξακολουθεί να υπάρχει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η απάντηση ήταν κρυστάλλινη, ναι. Και γι' αυτό λοιπόν, αν εδώ τώρα στα, του προπολογισμού ε, υπάρχουν κάποιε αποχρώσει, ε, αυτό δεν μ' αρέσει. Και αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ο πρώτο στόχο που, που έθιξε ο κύριο Μπρόκ, δηλαδή να υπάρχει μια εύρυθμα λειτουργούσα εξωτερική πολιτική. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ ο κύριο Κρίστοφερσον και συζητάει μαζί μα, όμω, αν αναφέρθηκε ήδη πώς θα, μας, ε, θα διαβουλευτούμε και θα συναποφασίσουμε και εμείς όταν μόνοι σας λέτε ότι το οργανόγραμμα είναι ανεπαρκέστατο ε, το σχέδιο αυτό των αποφάσεων δεν έχει καν παραρτήματα τότε και εμείς ε, πώς θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε μια σοβαρή διαδικασία διαβουλεύσεων. Γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτό που βλέπω στο οργανόγραμμα, όσο και αν είναι ανεπαρκές, για μένα δεν αρκεί για να έχουμε ένα μοντέλο αποτελεσματικής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ε, που προσφέρει το εξής, ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό Εθνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λάμπστορφ. Για δύο λεπτά ο κύριος Μπραντ, η κυρία Μπραντνα. Σύντομα να πω ε, τρία πράγματα. Κοιτάξτε, έχουμε ε, τα διάφορα ε, διακυβερνητικά στοιχεία, τα διάφορα στοιχεία και θέλω ε, να ξέρω κατά πόσον το μείγμα ε, θα είναι επιτυχημένο ή όχι και κατά πόσον όλα αυτά είναι διακυβερνητικά. Πρώτον, όσον αφορά τις αποστολές που μέχρι τώρα υπάγονται στη γραμματεία, οι αποστολές της κυρίας Άστον αλλά και του κυρίου Μπροκ θα είναι ξεχωριστές αυτές αυτό το αποφάσισαν τα κράτη-μέλη του 2009 και ρωτώ μήπως ε, παρόλα αυτά θα έχουμε ένα συγκερασμό προσωπικού, δηλαδή εκεί θα πάει προσωπικό ε, της Κομισιόν ή ε, το προσωπικό αυτό θα είναι τελείως ανεξάρτητο. Αν αυτό το κομμάτι παραμείνει πλήρως ε, ανεξάρτητο, τότε δεν θα μπορεί το προσωπικό αυτό να έχει χρήση του εργαλείου σταθερότητας. Γιατί στην περίπτωση αυτή πάμε σε διακυβερνητικές δομές και δεν αρκεί ε, στο τέλος να υπογράφει την επιταγή κάποιος που θα είναι από την Κομισιόν. Θέλω λοιπόν να μου το διευκρινίσετε αυτό. Κατόπιν αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας. Στην τελική πρόταση της κυρίας Άστον βλέπουμε ότι αυτή έχει και ε, δικαιώματα εκπροσώπησης. Αυτό μπορεί να ισχύει ε, σε κάποια χώρα όπου ο Υπουργός ε, να μπορεί να απολυθεί. Όμως ε, δεν μπορούμε να το ε, πετύχουμε αυτό και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με την κυρία Άστον. Δεν μπορούμε να την εκδιώξουμε. Άρα δηλαδή αυτό το θέλουμε. Ε, ποιος θα μπορεί να διορίζει τον Γενικό Γραμματέα, ποιος θα μπορεί να τον απολύει, γιατί ο Γενικός Γραμματέας να έχει τόσα πολλά δικαιώματα. Κατόπιν και αυτό το 1 τρίτο Ποιος θα ε, πληρώνει το, θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα κράτη-μέλη ή θα προέρχεται από τον ε, κοινοτικό προπλογισμό. Αν ε, πληρώνουν τα κράτη-μέλη είναι σαφέ σε ποιον θα είναι οι υπάλληλοι αφοσιωμένοι. Και αν τα χρήματα έρχονται από τον κοινοτικό προπλογισμό μπορείτε επιτέλους να μας πείτε πόσο θα κοστίσει αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ κύριε Μπράιτνερ. Ο κ. και έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ζήτησα το λόγο, αλλά εφόσον είμαι σκιώδη ηγητή, πρέπει να προβώ σε κάποια σχόλια. Αντίθετα από τη συνάδελφό μου, την κυρία Πράτνερ, η ομάδα μου βεβαίω που είναι μεταρρυθμιστική φύσεω και ευρωλεστική ομάδα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που πολλά στοιχεία τη νέα υπηρεσία θα είναι διεκβιντικής φύσεως υπό την αιγίδα του Συμβουλίου, κυρίω στον τομέα πολιτική προετοιμασία και υποστηρίξη ΚΕΠΑ και τη ΚΕΠΑ. Έχοντας ακούσει τη σημερινή συζήτηση, συμφωνώ με τον κύριο Λάμσδορφ, υπάρχει διάλογος μεταξύ κοφών ε, και σε ένα χρόνο όμως και παραπάνω, de facto, θα υπάρξει συνεννόηση όσον αφορά το πώς θα λειτουργεί όλη η υπηρεσία. Δα, κάποιοι ειδικοί με τον προπολογισμό θα πρέπει να αναλύσουν τον περιπλοκότατο προπολογισμό. Είναι πολύ περίπλοκο για του βουλευτέ. Ακόμα μετά από 10 χρόνια, εμεί οι βουλευτέ δεν το καταλαβαίνουμε και αν μέρει αυτό είναι σκόπιμο, το ώστε πραγματική εξουσία είναι στα χέρια εκείνων που κατανοούν τον προπολογισμό και ανακατεύονται με την εκτέλεσή του. Παρ' όλα αυτά, εν γέννη, η ομάδα μου υποστηρίζει πιο ευέλικτη εξωτερική υπηρεσία που επικεντρώνεται επί στρατηγικού σχεδιασμού σε τομεί όπω η ανάπτυξη αν αναγκαίων. Αυτό με εκπλήσει, λέγω ότι ήταν εκτό. Όμω επικρατεί όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, την ΚΕΠΑ. Με προβληματίζει το ότι είδα διάφορα οργανογράμματα που κυκλοφορούν. Και ποιος είναι ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα, που δεν είναι μεγάλος υποψήφιος από ό,τι μα λένε στον Βρετανικό τύπο. Κατά πόσο λοιπόν η PSC, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, που δεν την ξέρουμε καλά στο Κοινοβούλιο και είναι πολύ ισχυρή, κυρίως όσον αφορά τις στατιωτικές επιχειρήσεις, κατά πόσο ο μόνιμος πρόεδρός τους θα περνά μέσω της ιεραρχίας του Γενικού Γραμματέα ή αν θα είναι άμεσα υπόλογος στον ύπατο κόσοπο. Είστε κάτι με Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Ο κύριος Σάιρους Βόλσκι έχει το λόγο για ένα δίλεπτον. Ναι, ε, έπιασα κάποιον αφηρημένο. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα και δύο θέματα. Το... Θέλω μια διευκρίνηση. Πώς να το πω τον πρέσβη, πώς να τον αποκαλέσω. Γενικό διευθυντή. Όταν λέτε ότι ο κανονισμός προσωπικού θα είναι ανοιχτός για κάθε θεσμικό όργανο, εννοείται και για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όχι δύο θέματα τονίσω. Σαν Κοινοβούλιο θέλουμε ισχυρή εξωτερική πολιτική και προφανώς ισχυρό εργαλείο για να το πραγματοποιήσουμε. Δύο ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα ο πολιτικός έλεγχος αναφέρθηκε και το πρόβλημα είναι ότι δεν θα υπάρχει αρκετός πολιτικός έλεγχος όπως θα θέλαμε αν η Λέβη Άστον ε, εκτελεί τέσσερα καθήκοντα και δεν θα έχει βοηθούς, αναπληρωτές. Πώς θα εκπροσωπείτε σε πολιτικό επίπεδο το κοινοβούλιο, κάτι που απαιτείται. Γνωστά τα επιχειρήματα, απλώς θέλω να το θέσω το ζήτημα. Τρίτο, νομιμότητα. Η υπηρεσία πρέπει να γίνει δεκτή από μόνη της, από όλου τους πολίτες των κρατών μελών. Άρα χρειάζεται η γεωγραφική αντιπροσωπευτικό τη. Ερώτηση. Πόσο αντιπροσωπευτική θα είναι η ύπατη εκπρόσωπος αν η υπηρεσία τη δεν είναι αντιπροσωπευτική. Η γεωγραφική ισορροπία χρειάζεται, η γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, να αισθανθούν ότι τους ανήκει αυτή η υπηρεσία. Και όλοι οι πολίτε των κρατών μελών, βορρά, νότων, Ανατολή και Δύσεω, να συμμετέχουν, ότι να θεωρούν ότι εκπροσωπούνται. Άρα, αρμοδιώτης ε, δεν μπορεί να θεωρείται ως γεωγραφικά ουδέτερη, Διαφορετικά χρειάζονται ενδεικτικοί στόχοι για όλους τους υπηκόους. Ενδεικτική προσέγγιση και κάποια προσωρινή πρόβλεψη βάσει του κανονισμού 401 του 2004 του Συμβουλίου όσον αφορά την αρχική κατέθεση που ακολουθηθεί. Ευχαριστώ κύριε Σάιλος Βόλσκι. Κύριος Βόμποντα έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Well, um, I agree with the... Συμφωνώ με τον κύριο Κριστόφερσον. Είπε ότι χρειάζεται ευελιξία για να μάθουμε μέσω της εμπειρίας. Βέβαια κάποια στοιχεία όμως θα πρέπει να καθοριστούν. Ένα από τα στοιχεία όσον αφορά τον προπολογισμό ε, πρέπει να αναλυθεί. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές εμείς σοσιαλδημοκράτες. Δεν είναι μόνο το θέμα της δομής, αλλά θα πρέπει να ελέγχουμε τον προπολογισμό και να χορηγείται απαλλαγή. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Αν υπάρχουν εγγυήσει με την παρούσα πρόταση, γι' αυτό καλώς. Διαφορετικά θα πρέπει να βρούμε άλλη λύση για το προσωπικό. Και μιλώ εκ μέρους του κύριου Ράπκα που είναι εισηγητής. Δεν είμαστε σίγουροι ότι τα μέτρα εγγυώνται ότι θα υπάρχει από μία πηγή το προσωπικό που θα είναι εκεί. Αν είναι από το Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα κράτη-μέλη, θα πρέπει οι πολίτε και άλλε χώρε όλοι να ξέρουν ξεκάθαρα ότι είναι ένα το προσωπικό, ενίο το προσωπικό και θα πρέπει να ακολουθεί τη γραμμή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και όχι εθνική γραμμή. Συμπεριλαμβανομένων και των ευθυνών ε, σε περίπτωση λαθών. Και πιστέψει κάποιο στο Υπουργείο του στη χώρα του. Αν κάτι πάει στραβά θα φέρει την ευθύνη αυτός για τα λάθη του. Ελπίζουμε όμως να μην ε, συμβεί κάτι τέτοιο. Για το Γενικό Γραμματέα. Είναι διοικητική θέση κατά την άποψή μας. Και η κυρία Άστον, η ύπατη εκπρόσωπος θα πρέπει να αποφασίσει για την προσωπικότητα. Χρειαζόμαστε πολιτική εκπροσώπηση. Δεν μιλώ για τους αναπληρωτές γιατί είναι κάπως παραπλανητικό και δεν βασίζεται στη συνθήκη. Αν έχουμε ύπατο εκπρόσωπο βάση του άρθρου 33, ίσως ύπατος εκπρόσωπος για επικοινωνία, για διοργανικές σχέσεις, όπως έχουμε αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα είναι αυτός ή αυτή. Χρειαζόμαστε προσωπικότητα για επαφές με το Κοινοβούλιο. Σκεφτείτε και αυτό. Εμείς σαν ομάδα είμαστε πραγματιστές, κάποια στοιχεία όμως πρέπει να καθοριστούν. Ευχαριστούμε και ολοκληρώνει το δεύτερο γύρο των παρεμβάσεων η κυρία Γιαννάκου. Για δύο λεπτά παρακαλώ κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τι θέλουμε να δημιουργήσουμε, αυτό που επί χρόνια όλοι ζητούσαμε, μια πραγματική εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ε, η Λέιδη Άστον βεβαίως είναι ως επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά στην ουσία πρέπει να εκπροσωπεί την Ένωση και η Ένωση περιλαμβάνει και το Κοινοβούλιο. Επομένως όσα ελέγχθησαν από την προηγούμενη φορά, δηλαδή να υπόκειται στην απαλλαγή του Κοινοβουλίου και όλα τα σχετικά, αυτό πρέπει να ισχύσει. Άλλα ζητήματα όπως είναι η γεωγραφική κατανομή κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς εξασφαλίζουν το να ανατραπεί από την αρχή της αυτή η προσπάθεια για δημιουργία εξωτερικής πολιτικής αν δημιουργηθούν προβλήματα με ορισμένες χώρες απόκλησης από κάποιες γενικές αρχές ή ασύμβατες καταστάσεις με τα συμφέροντα ορισμένων χωρών θα υπάρξει πρόβλημα στην αρχή. Γι' αυτό και η γεωγραφική κατανομή και ο σεβασμός αυτής της έννοιας νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία καθώς και η δημιουργία μιας ομάδος που θα έχει εμπειρία και θα προέρχεται και από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο, αλλά και ανεξάρτητοι ικανοί άνθρωποι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη στελέχωση αυτής της ομάδος. Ευχαριστούμε την κυρία Γιαννάκου. Τώρα λοιπόν ε, θα δώσουμε το λόγο στους ε, φιλοξενούμενους μας με την ίδια σειρά όπως και πριν. Ε, ξεκινάμε ε, με τον κύριο Κρίστοφερσεν. Να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Λάμπστορ. Πρέπει λοιπόν, όπως σας είπαμε, να περιμένουμε τρεις εβδομάδες ε, γιατί θα έρθει το παράρτημα και αυτό σίγουρα θα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την αξιολόγηση του συστήματος. Τώρα, όσον αφορά στο οργανόγραμμα, εγώ ε, εξακολουθώ να τάσσομαι υπέρ της ευελιξίας. Ε, έχουμε τη μονάδα που επιθυμούμε, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην τραβήξουμε πολλές γραμμές ανάμεσα σε αυτή τη μονάδα γιατί θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις καταστάσεις που θα ανακύψουν και θα πρέπει, είπατε, να υπάρχει ένας μετριοπαθής υπουργός εξωτερικών και ένας ε, που γνωρίζω πολύ καλά ε, δεν έχει τραβήξει καθόλου γραμμές ε, στην υπηρεσία του. Η μετακίνηση γίνεται ανάλογα με, τις, με τα γεγονότα και την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί. Και φτάνω λοιπόν στα ερωτήματα που ετέθησαν σχετικά με τον Γενικό Γραμματέα. Πρώτα απ' όλα Επιτρέψτε μου να καταστήσω σαφές ότι όταν λέμε ότι ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να εκπροσωπεί την υπηρεσία, δεν εννοούμε πολιτική εκπροσώπηση. Αν θέλετε να προσθέσετε να εκπροσωπεί την υπηρεσία στο επίπεδό του, να προσθέσετε δηλαδή το at his level, στο επίπεδό του, μπορείτε να το προσθέσετε Σαφώς κανένα πρόβλημα. Εγώ όμως δεν συμφωνώ με εκείνους που λένε ότι δεν χρειαζόμαστε ισχυρό γενικό γραμματέα. Εγώ διαφωνώ, χρειαζόμαστε ισχυρό γενικό γραμματέα γιατί ένα, ένας από τους βασικότερους ρόλους που θα παίξει είναι ο ρόλος του συντονισμού της ε, εξωτερικής πολιτικής, ε, κάτι το οποίο αφορά την κυρία Άστον και προϋποθέτει το συντονισμό με την Επιτροπή, με την ε, Γραμματεία του Συμβουλίου να είναι ένα ισχυρό πρόσωπο. Γι' αυτό λοιπόν είναι ε, εφησυχασμός για την, είπα το εκπρόσωπο, να έχει κάποιον που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας ε, είναι πολύ σημαντικός στο να διασφαλίζει το συντονισμό στο εσωτερικό υπάρχει σαφώς ανάγκη ε, συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντονισμός ανάμεσα στις ε, αποστολές ε, ΚΕΠΑ, συντονισμός ανάμεσα σε πολλές άλλες περιπτώσεις και όλα αυτά πρέπει να τα κάνει ο Γενικός Γραμματέας ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος ε, θα διασφαλίζει ότι ε, το οργανόγραμμα και η οργάνωση λειτουργεί αποτελεσματικά. Και σας παρακαλώ να ξεχάσετε όλα τα ονόματα που αναφέρονται στον τύπο. Ξέρετε, μιλάτε εκτό μικροφώνου, γυρίζει ο μιλητή και ξεχνάει το μικρόφωνο. Αλλά για να ακούν διερμηνεί πρέπει να μιλάτε στο μικρόφωνο, λέει και ο πρόεδρο. Λοιπόν, ξεχάστε όλα αυτά τα ονόματα που κυκλοφορούν. Όλοι οι ανώτατοι διορισμοί συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Γραμματέα θα, είναι, θα περάσουν μέσα από διαδικασία επιλογής. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περάσουν μέσα από την ίδια διαδικασία επιλογής ε, ε, και αυτό ισχύει για όλους τους επικεφαλείς αντιπροσωπιών. Σήμερα, για να μετεφερθεί κάποιος ε, από την Επιτροπή σε εξωτερική θέση, αυτό θα γίνει με το νέο σύστημα. Όλες οι θέσεις θα επάγονται στο νέο σύστημα. δεν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σβόμποντα για την ευελιξία του και θα ήθελα να επαναλάβω ότι αν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το τι έχει υποσχεθεί η κυρία Άστον ότι θα υπάρχει η ίδια διαδικασία προϋπολογισμού και απαλλαγής ε, αν υπάρχει οποιαδήποτε εμφολία τότε να αλλάξετε το κείμενο γιατί εμεί αυτό επιθυμούμε να μην υπάρχει ε, καμία αμφιβολία επί του στόχου ε, κατά πόσον τα καταφέραμε δεν το γνωρίζω αλλά εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει οποιαδήποτε εμφολία μπορεί να υπάρξει και κάποια αλλαγή ευχαριστούμε το λόγο έχει ο κ. Ζανζουάν Ζουάν Πρόεδρε, θα είμαι λακωνικότατο, διότι νομίζω ότι έδωσα όλε τι αναγκαίε διευκρινήσει. Ένα σημείο μόνο. Προπολογισμό θα καλύπτει αυτός σύνολο διοικητικών δαπανών και, ε, και την αμοιβή των προσωρινών υπαλλήλων, τους διπλωμάτες δηλαδή με άλλα λόγια, που θα εργάζονται εντός της εξωτερικής υπηρεσίας. Θα το πω διαφορετικά ότι θα υπάρχει ισότητα μεταξύ όλων εντός αυτής της υπηρεσίας. Κατά λοιπά, νομίζω ότι απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζωάν, κύριε Σούκα. Θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είπε ο συνάδελφος. Επιπλέον, οι εθνικοί διπλωμάτες όχι μόνο θα πληρώνονται από τον κοινοτικό προπολογισμό, αλλά δεν επιτρέπεται να δεχθούν η πληρωμή από οποιαδήποτε άλλη πηγή εκτός του θεσμικού αυτοργάνου. Δεν θα έχουν άλλη πληρωμή, άλλη αμοιβή από τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Ένα δεύτερο ερώτημα που ετέθη είναι σε ποιο βαθμό οι υπάλληλοι, τα μέλη άλλων θεσμικών οργάνων θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Αυτό που είπαμε είναι ότι θα κάνουμε διάκριση μεταξύ της αρχικής φάσης όπου θα έχει κανείς μόνο υπαλλήλου που θα προέρχονται από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κατημέλη και κατόπιν αφού θα λήξει αυτή η αρχική φάση τότε η πρόσβαση στην, εξωτερική υπηρεσία, ε, στην υπηρεσία εξωτερική δράση ε, θα είναι η υπηρεσία αυτή ανοιχτή σε υπαλλήλου από όλα τα θεσμικά όργανα. Το τελευταίο θέμα που ετέθη, σε ποιο βαθμό οι προσωρινοί υπάλληλοι όταν επιστρέψουν στα κράτη-μέλη θα εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για τι δράσει του, για τι πράξει του στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Βέβαια είναι ένα θέμα που υπάρχει με όλου του προσωρινού υπαλλήλου, δεν είναι νέο πρόβλημα. Το είχαμε πει σειρά ετών όλα δεσμικά όργανα το πρόβλημα, σε ποιο βαθμό, τι εξουσίε έχουμε έναντι των προσωρινών υπαλλήλων τη στιγμή που θα αποχωρήσουν. Αλλά εφόσον υπάρχουν πάντα οικονομικέ σχέσει, συντεξιωτικά δικαιώματα που αποκτώνται και άλλα συναφή, νομίζω ότι έχουμε κάποια εξουσία πάνω του, Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο το θέμα και βλέπω ότι υπάρχει ευαισθησία στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σούκα. Τελευταίος γύρος, δύο λεπτά για τον κύριο Νταφ. Πρόεδρε, ο κύριος, κύριε Κριστόφερσεν. Θέλω να επανέλθω στο ζήτημα των αναπληρωτών της ε, κυρίας Άστον εμάς είναι πάρα πολύ βασικό, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το ποιος θα συνομιλεί με το Κοινοβούλιο. Αλλά το θέμα είναι το τι θα γίνεται σε υπουργικό επίπεδο. και όσον αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Γιατί είπαμε ότι δεν ήταν να έχουμε την Προεδρία και τη Γενική Γραμματεία που δεν μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο όπως είστε και οπότε σας παρακαλώ να με ενημερώσετε σε αυτό το θέμα ε, με ενδιαφέρει πολύ. Κατά δεύτερο λόγο νομίζω ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα ένα πρόβλημα χρονοδιαγράμματος, χρονισμού αν θέλετε ε, ε, γιατί όσον αφορά την πρόοδο στα σχετικά ζητήματα κάπω έχει χαθεί ο δυναμισμό η δυναμική οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα και θα πρέπει τώρα να προχωρήσουμε σε μια διοργανική συμφωνία κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι μια συζήτηση τετραμερής και να συμμετέχει σε αυτό και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μια που είναι κομβικός ο του σε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ κύριε Νταφ. Κύριε Σεβερίν έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε όσον αφορά την ερμηνεία της συνθήκης. Δηλαδή με, ρητά, ρητό τρόπο ή εννοείται ότι η συνθήκη μας ζητά να κάνουμε τα δέοντα ούτως ώστε να έχουμε μια συνεκτική, πλήρη και αποδοτική και δραστήρια εξωτερική δράση. Ενεργό εξωτερική δράση. Αυτός ο στόχος νομίζω ότι η συνθήκη μας επιτρέπει να βρούμε η αδίποτε λύση για να πετύχουμε το στόχο. Διότι οποιοδήποτε εμπειρογνώμονας για θέματα νομικά θα σας πει ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε, να, δούμε εμείς, να έχουμε μια συνθήκη που θέτει ανέφικτους στόχους. Αν περί αυτού πρόκειται, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές δρα... ε, πτυχές και σύμφωνα με τη συνθήκη υπάρχουν διάφορα κέντρα αρμοδιοτήτων. Και το ερώτημα που θέτω στους ε, φιλοξενούμενους μας, ε, καταρχάς, πώς, πείτε μας μια διατύπωση που να μας επιτρέπει να εξηγήσουμε στους ψηφοφόρους μας, στους Ευρωπαίους πολίτες μας, ότι μπορούμε να έχουμε στρατηγική εξωτερικής δράσεως, μια <coughs> στρατηγική για την ΚΕΠΑ, η οποία να είναι συνεκτική και ότι ο μηχανισμός που δημιουργούμε μέσω αυτής της υπηρεσίας θα μας επιτρέπει να καθορίσουμε μια τέτοια πολιτική. Δεύτερον, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες μας ότι τα δημοσιονομικά μέσα που χρειάζονται για να χρηματοδοτήσουμε μια τέτοια πολιτική και χωρίς αυτά τα εργαλεία δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η πολιτική και αυτά ε, σχεδιάζονται με έναν τρόπο που εξασφαλίζει συνοχή δημοσιονομική ε, και τη σχετική συνοχή της πολιτικής. Πώς εξηγούμε ότι όσον αφορά το προσωπικό μπορούμε να ισορροπήσουμε τη γεωγραφική εκπροσώπηση Κάτι που τόνισε ο κύριος Σάιρους Βόλσκι. Με την ε, ευρωπαϊκή ταυτότητα και πιστότητα την ευρωπαϊκή του να, να ανήκουν αυτά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Σεβερίν. Λούνατσεκ, για δύο λεπτά είναι το επόμενο όνομα. Κυρία Λούνατσεκ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ να συνεχίσω αυτά τα οποία είπε η κυρία Σούκα πριν από λίγο όσον αφορά το ζήτημα του τι γίνεται όταν έχουμε τους ε, επικεφαλείς των αντιπροσωπιών οι οποίοι επανέρχονται στη χώρα τους ε, αναλαμβάνουν κάποια θέση πρέσβεως. Τι γίνεται εδώ όταν έχουμε κάποιο είδους ε, προβλήματα. Βεβαίω και έχουν ασυλία διπλωματική. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνετε. Άρα χρειάζεται να κλείσει κάποια συμφωνία με τα κρατημέλη και να υπάρξουν διαβεβαιώσει ότι σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάτι αντικανονικό να αφορά την υπηρεσία εξωτερική δράση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να στραφεί εναντίον του. Οπότε παρακαλώ σκεφτείτε και αυτό μέσα μετά που είπα ότι θα σκεφτείτε. Θα πρέπει να συναφεί κάποια συμφωνία με τα κράτη από αυτού. Τώρα κάτι άλλο το οποίο επίση είναι σημαντικό για όλου μα. Ποιο πρόκειται να ορίσει τον ε, γενικό. Ο κύριος Κριστόφος μας είπε κάτι για τη ε, διαδικασία της επιλογής που θα ακολουθεί η κλασική διαδικασία για τις ψηλές θέσεις. Ποιοι θα τους επιλέξουν. Και όλα αυτά μας βρίσκουν Αυτοί οι οποίοι θα αποσπώνται από τα κράτη-μέλη. Θα πληρώνονται από τον κοινωτικό προπολογισμό. Πόσο? Όσοι θα έρχονται εδώ με απόσπαση. Τι θα γίνει, αυτό έχει σημασία για μας. Κάτι άλλο για τον προπολογισμό επίσης. Σε, συμφωνεί με αυτά τα οποία είπε για την ΚΕΠΑ ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ναι, εμείς όντως θέλουμε να έχουμε ε, όντως κάποια έξτρα κονδύλια. Νομίζω θα κάνει πιο εύκολο το έργο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Πορέμπα το επόμενο όνομα για δύο λεπτά. κ. Πορέμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα απευθυνόμενο προς τον κύριο Κριστόφερσον, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, στο νέο αυτό σώμα των διπλωματών, στο στελέχη αυτά, ετίθετο το θέμα του εγγυημένου 50% εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι γνωστό ότι τα νέα κράτη-μέλη δεν έχουν αρπαρκή εκπροσώπηση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα και θεωρώ ότι θα μπορούσαν να θα μπορούσαν στο σύστημα να υπάρχει κάποια διάκριση έτσι όσο έχει κατά των νέων κρατών μελών όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Είπατε εκπρόσωπος Βαρόνι Άστον θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στον εξωκόσμο. Ε, πώς μπορεί κανείς να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στον έξω κόσμο, στην τομέα της εξωτερικής πολιτικής, αν υπάρχει ανισορροπία εσωτερική όσον αφορά το προσωπικό. Αυτό δεν θα έχει συνέπειες όσον αφορά την αλληλεγγύη και την εθνική και γεωγραφική ισορροπία. Είναι σημαντικά στοιχεία. Ακόμα αν αυτό σημαίνει και ποσοστώσεις που θα υπάρχουν η ισορροπία στην, ε, στις θέσεις εργασίας θα είναι κάτι πολύ σημαντικό αν θέλουμε η υπηρεσία εξωτερικής δράσεως ε, να είναι αμερόληπτη. Και δεν είναι καλό να υπάρχουν ανισορροπίες και διακρίσεις ε, γενεί στο σύστημα αυτής εξ αρχής. Ευχαριστώ κύριε Πορέμπα. Ο κ. Μίλαν Μόν έχει το λόγο για δύο λεπτά. Θα είμαι πολύ σύντομος πρόεδρε γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σωστό το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια γεωγραφική ισορροπία, να διασφαλιστεί αυτό ακριβώ όπω ισχύει και τώρα και του τόνισαν συνάδελφοι. Επίση θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσει να ισχύει το ότι αυτό το εξάμεινο θα υπάρξει η έγκριση ακριβώ όπω αρχικά είχε προβλεφθεί. Θα ήθελα να μου το ξεκαθαρίσετε αυτό. Επίση σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όσο μα ξεκαθαρίσατε όσον αφορά του υπαλλήλου που έρχονται από τα κράτη-μέλη. Μιλήσαμε για 600-700 από την Κομισιόν, 50 ε, είπατε από το Κοινοβούλιο και περίπου 200 στρατιωτικοί. Τελικά όμως για πέστε μας, τι, τι, τι, τι ισχύει, τουλάχιστον για τα κράτη-μέλη. Τώρα, μια διευκρίνηση. Εάν κατάλαβα καλά, η, η, η πρόσληψη αυτών που θα είναι από τα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι σωστό, γιατί νομίζω ότι θα, θα δώσουν κάποια νέα πνοή και ξέρουν και τα θέματα, ότι θα είναι λοιπόν ο ορισμός τους θα είναι προσωρινός. Τι γίνεται τώρα με τους ε, ε, επιτρόπους της Κομισιόν, αυτή θα είναι μόνιμη ή προσωρινοί, γιατί τότε θα έχουμε μια ανομοιογένεια μεταξύ των μεν και των δε. Ευχαριστώ κύριε Μίλαν Μον. Βαϊντέρε το επόμενο όνομα για δύο λεπτά. Κυρία Βαϊντέρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν ήδη και ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια θέματα που αφορούν το προσωπικό. Όπως βλέπω τα πράγματα, αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα πρέπει να είναι ισχυρός ε, φορέας που θα πραγματοποιεί ισχυρή εξωτερική πολιτική. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω με την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Γαλλικού τύπου, διότι είχαμε πολλούς θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που κινούνται μέσω του προσωπικού και είναι κατά αυτού οι πολίτες. Θέλουν καλύτερη εκπροσώπηση ε, σε αυτά τα θεσμικά όργανα. Και είπατε επίσης ότι πρέπει να λησμονήσουμε όλα αυτά που αναφέρονται στον τύπο για την επιλογή του Γενικού Γραμματέα. Και το θέμα είναι πώς θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Και πόσο σίγουρο μπορεί να είμαστε... Τα παιδιά να είναι ξανά Γάλλος ε, μετά από αυτή τη διαδικασία προσδίψεως ο, ο Γενικός Γραμματέας. Το θέμα που ετέθη από συναδέλφο, το συνάδελφο Σάριος Βόλς και την κυρία Γιαννάκου Μπορέμπα για τη γεωγραφική εκπροσώπηση, γεωγραφικές αρχές. Δεν είδα να υπάρχει αυτή η γεωγραφική εκπροσώπηση. Και αυτή η έννοια της ιδιοκτησίας είναι κάτι πολύ σημαντικό στην εξωτερική υπηρεσία. Διαφορετικά ε, θέλουμε αυτός ο θεσμός ε, εγώ είμαι από, από μικρή χώρα, από τη δηλαδή, α, και θέλω να δω και διπλά σε εκπροσώπηση. Και αν, ε, θα πρέπει οι χώρες μας, οι μικρές μας χώρες να εκπροσωπούνται. Δεν εκπροσωπούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν ακολουθηθεί λάθος προσέγγιση θα εκπροσωπούνται και σε αυτό το νέο φορέα. Και δεν θέλουμε άλλο ένα γραφικό θεσμό. Eh, Υπάρχει μια παρέβαση του κυρίου Μπράτνερ, τη κυρία Μπράτνερ, για τον κανονισμό. Κοιτάξτε, μία ερώτηση δεν απαντήθηκε και είναι πολύ σημαντική για μας, δηλαδή κατά πόσον στη διαχείριση των ε, κρίσεων θα προσληφθεί ε, προσωπικό ε, και από άλλες διευθύνσεις και όχι μόνο από τις Γενικές Διευθύνσεις των Κρατών Μελών θα απαντήσετε μετά, όταν ε, θα απαντήσουν ε, οι φιλοξενούμενοι μας. Αντρίκινεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, αλλά η δική μου ερώτηση και αυτή αφορά ε, στην γεωγραφική εκπροσώπηση και θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μόνο σε αυτό το θέμα εκεί που γίνεται για τον ε, διορισμό ανώτατων ε, στελεχών. Εγώ είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι η νομοποίηση της υπηρεσίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την γεωγραφική εκπροσώπηση ε, του προσωπικού. Έτσι λοιπόν αυτό που έχουμε ε, στο έγγραφο μπροστά μας, ε, το οποίο προετοίμασε ο συνάδελφός μας, ο κύριος, οι κύριοι Μπροκ και Φερχόφστατ, υπάρχουν δύο εναλλακτικέ λύσεις όσον αφορά ε, στην διαδικασία των διορισμών. Ε, η διαδικασία είναι ότι ο διορισμός μπορεί να γίνει ε, και μέσα από τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών. Άρα δηλαδή πρέπει να επιμεριστεί η αρμοδιότητα ε, για την υπηρεσία αυτή ανάμεσα στην Κομισιόν και το Συμβούλιο και κατόπιν θα πρέπει να υπάρχει ίσως ε, μια επιτροπή επιλογής ε, όπου ε, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους της Κομισιόν και του Συμβουλίου και των κρατών μελών. Οι αρχές που αναφέρονται εδώ είναι οι αρχές της, των προσόντων και της ε, εκπροσώπησης εις εκπροσώπησης γεωγραφικής και των δύο φύλων. Ε, επιμένω ε, σε αυτό που είπε ο κύριος Βολσκι στο θέμα των προσόντων και της γεωγραφικής εκπροσώπησης και εκπροσώπησης των δύο φυλών. Θα εκτιμούσα πάρα πολύ ο κύριος Κριστόφασταν και οι συναδελφοί του να σχολιάσουν αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κλείνει με μια σύντομη παρέμβαση ο κύριος ε, Κόμπατσεφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε, θα είμαι πολύ σύντομος. Για τον κανονικό προσωπικού, αυτή η αρχική φάση κίνησης της διπλωματικής υπηρεσίας πόσο θα κρατήσει χρονικά, Δεύτερο, δεν επαναλαμβάνω αυτό που είπαν οι συνάδελφοι για τη γεωγραφική ισορροπία, αλλά για τη μέθοδο. Μία μέθοδος θα μπορούσε να είναι να χρησιμοποιήσουμε τον κανονισμό 401 του 2004 ε, για την εκπροσώπηση των κρατών μελών. Ξέρουμε ότι στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποεκπροσωπούνται τα νέα κράτη-μέλη. Ε, θα επαναληφθεί η προσέγγιση που ακολουθήθηκε το 2004. Ευχαριστώ κύριε Κόβατσεφ. Ο κύριος Κρίστιανσεν για 3-4 λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πολλές ερωτήσεις ε, να απαντηθούν σε 4 λεπτά. Καταρχάς, το θέμα των ε, πολιτικών εκπροσώπων. Αυτό είναι κάτι που ετέθη επιτάπητος και δεν θα χαθεί. Θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα σημαντικά θέματα που θα συζητηθεί στο φόρουμ. Και συμφωνώ με τον κύριο Νταφ που το ταχύτερο δυνατόν θα πρέπει να συσταθεί και να συζητήσει. Είναι μια ιδέα πολύ ελκυστική, αλλά είναι και περίπλοκη. Και υπάρχουν και δεχόμενοι τομείς σύγκρουσης. Όχι τόσο πολύ με το Συμβούλιο, αλλά περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έλεγα. Θα υπάρξει κάποιος ε, αντιεπίτροπος του ΣΥΠΗΝ, εκπρόσωπος του, του Επιτρόπου, απεσταλμένος εκπρόσωπος και αν ασχοληθεί αυτός ο εκπρόσωπος με θέματα που είναι ευθύνη και του Επιτρόπου Ανάπτυξης, Φερρυπίν, εμείς είμαστε έτοιμοι προς συζήτηση αυτών. Δεν είναι δουλειά μου να μαντέψω τι θα κάνουν τα άλλα θεσμικά όργανα και τι θα πούν. Για αυτό που είπε Άντριο Ντόφ, για παράλληλη συζήτηση. στην τετράπλευρη αυτή μορφή συζητήσεων για τον πολιτικό έλεγχο. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Το ταχύτερο δυνατόν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό μπορώ να πω από την πλευρά μου. Ετέθησαν πολλά ερωτήματα σχετικά με το προσωπικό, σχετικά με τη γεωγραφική ισορροπία. Να προσπαθήσω λοιπόν να καλύψω τα διάφορα θέματα. Στην προσωπική μου ζωή Δύο φορέ ήμουν αποσόλιο υπαλλήλο. 14 χρόνια στην Γραμματεία του Συμβουλίου και 4 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι θεωρούσα τον εαυτό μου πλήρη υπάλληλο της κοινότητας κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου η ιδέα ότι κατά κάποιο τρόπο ανήκει στην εθνική σου δίκηση ε, δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο αισθανόμουν εγώ τουλάχιστον κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Στο σύστημα θεωρήσαμε μια κανονική περίοδο για το προσωπικό αποσπασμένο στην υπηρεσία 8 χρόνια, 2 επί 4. Και αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να δεχτούν αυτά τα άτομα αν θέλουν να επιστρέψουν. Αυτοί είναι οι κανόνες ε, που αναφέρουν στην απόφαση. Μετά την οκταετία, σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού, έχουμε εξαίρεση και δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να δεχτούν εκ νέου το προσωπικό. Όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία, αν υπάρχει ένα μήνυμα που ακούστηκε πολύ ηχηρά κατά τη διάρκεια της συζητήσεως ευθύς εξ αρχής είναι η απογοήτευση όσον αφορά τα νέα κράτη-μέλη. Αυτό που αισθάνονται τα νέα κράτη-μέλη όσον αφορά τη γεωγραφική εκπροσώπηση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ελήφθη το μήνυμα. Και γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι αν αυτή η ισορροπία δεν υπάρξει θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποιου μηχανισμούς για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Θα υπάρχει ετήσια έκθεση από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο, θα υπάρξει συμβουλευτική επιτροπή για διορισμό, όπου τα κράτη-μέλη θα συμμετέχουν στη διαδικασία διορισμών και θα μπορεί επίσης να συστήνει λύσεις στον ύπατο εκπρόσωπο αν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία. Τέλος, μάλλον στο Γενικό Γραμματέα για μια ακόμη φορά. Καταρχήν, η διαδικασία διορισμού του Γενικού Γραμματέως θα είναι η ίδια όπως και για τις άλλες θέσεις ανατέρων στελεχών. Θα δημοσιεύεται η θέση, θα υπάρχει επιτροπή επιλογής που θα κατατίζει ένα κατάλογο ε, και ο ύπατος εκπρόσωπος, η ύπατη εκπρόσωπος θα επιλέγει αυτό το κατάλογο και στην Επιτροπή Επιλογή θα υπάρχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών τη Γραμματεία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίω των συναφών φορέων. Στην κυρία Μπράτνερ, συγγνώμη που δεν απάντησα στο ερώτημα στην προηγούμενη φορά. Όσον αφορά την ΚΕΠΑ, υπάρχει έλλειψη προσωπικού για την ώρα. Λείπει το πολιτικό προσωπικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί στατιωτικοί για την ώρα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε και άλλα πολιτικά στελέχη, πολίτες και θα θέλαμε ε, και πολύ να έχουμε εκπροσώπους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ και λυπάμαι αν δεν απάντησα σε κάποιες ερωτήσεις. Κοιτάξτε, υπήρχαν κάποια όρια χρονικά. Η κυρία Σούκα έχει κάποιες απαντήσεις να δώσει. Ναι. Πρώτα απ' όλα είπατε πόσο θα πληρώνονται οι εθνικοί διπλωμάτες, θα είναι προσωρινοί υπάλληλοι, άρα θα πληρώνονται σύμφωνα το μισθό που συνδέεται με το βαθμό της θέσης που θα κατέχουν. Δεύτερο ερώτημα που ετέθη ήταν τι θα γίνει με τους υπαλλήλου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θα αποσπώνται στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Όχι, θα ε, μετακινούνται, θα μεταφέρονται και θα είναι υπάλληλοι τη επίτροπή. Δεν υπάρχει θέμα απόσπασης ή κάτι άλλο, θα είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μεταφερθούν, θα γίνουν υπάλληλοι της υπηρεσίας αυτής. Άλλο ερώτημα ήταν η αρχική φάση πόσο θα κρατήσει. μεταφερθουν θα γινουν υπαλληλοι τη υπηρεσία αυτή. αλλο ερωτημα ηταν η αρχικη φαση όριο στο, στο κείμενο που προτείνουμε, 1η Ιουλίου 2013. Τελευταίο ερώτημα αφορούσε την υποεκπροσώπηση των κατών μελών, κυρίως των νέων κατών μελών. Και αν κατάλαβα σωστά το ερώτημα, το θέμα ήταν σε ποιο βαθμό θα ήμασταν πρόθυμοι να παρατείνουμε τον κανονισμό για παρέκκληση του 2004, ώστε να προσλάβουμε στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης υπηκόους των νέων κατών μελών. Πιστεύω ότι αυτό είναι το ερώτημα που θέτατε και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτό το θέμα, να εξεταστεί. Κύριε Κριστόφερσεν, ίσως εσείς έχετε κάτι να πείτε. Υπήρχε και ένα θέμα για διπλωματική κινητικότητα. Ακινησία μάλλον ήρθε. Πώς να το πω. Ασυλία, ασυλία. Ασυλία, η διπλωματική ασυλία. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ήμουν και δίπλωμάτης στην καριέρα μου. Σαν διπλωμάτης έχεις ασυλία για τα καθήκοντα που ασκείς. Δεν σου παρέχεται ασυλία για άλλα πράγματα που έχεις κάνει κατά το παρελθόν σου. Αν έχεις λογαριασμούς να ξεκαθαρίσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διπλωματική ασυλία της Βορείας Κορέας δεν σε σώζει από το να πρέπει να πληρώσεις το... τα σπασμένα. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. Άλλα πέντε λεπτά έχουμε το πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για να ολοκληρωθεί το πλαίσιο με την τελική απάντηση του εισηγητού μας, του κυρίου Μπροκ. Έχετε το λόγο κυρία Μπροκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα που δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη Βόρεια Κορέα σαν ασπίδα μας. Κρίμα, κρίμα. Δεν έχει μείνει καμιά ελπίδα πια και αυτό ισχύει για τα μέλη βέβαια. Επιτρέψτε μου λοιπόν κάποιες ε, παρατηρήσεις. Εγώ νομίζω ότι σε ορισμένα σημεία πράγματι προέκυψε ε, ε, μεγαλύτερη διαφάνεια σε θέματα απαλλαγή στον δημοσιονομικό κανονισμό, στην πρόταση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει βέβαια να επανεξετάσουμε, να δούμε κατά πόσον ευσταθεί. Θεωρώ ότι το θέμα της πολιτικής εκπροσώπησης τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο όσο και το προσωπικό. Επ' αυτού δεν εξαντλήθηκε η συζήτηση. Και νομίζω αυτό φάνηκε με απόλυτη σαφήνεια. Πρέπει λοιπόν να είναι σαφές ότι οφείλουμε να κάνουμε σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στο ε, ποιες είναι οι συμφωνίες ανάμεσα στους θεσμούς και πού ακριβώς, ακριβώς υπάρχουν στοιχεία πρακτικής ε, συνεργασίας. συνεργασία ανάμεσα στην ΕΠΑ το εκπρόσωπο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ε, τις επόμενες εβδομάδες ε, θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να εξετάσουμε αυτά τα θέματα και ελπίζω να μην πει τελικά η ΕΠΑ εκπρόσωπος ότι στους τομείς αυτούς δεν θα κάνει τίποτα αυτόνομα γιατί τότε θα προκύψει πραγματικά πρόβλημα και εδώ εμπίπτει και το θέμα της πολιτικής εκπροσώπησης. Στήξαμε το οργανόγραμμα με τους δύο επιτρόπους και τους ε, δύο αναπληρωτές. Επ' αυτού ακόμα δεν ελέγχθη τίποτα τόσο σημαντικό. Αλλά ε, και από πλευράς ε, Κοινοβουλίου το θέμα είναι ότι έχει σημασία να υπάρχει σωστή πολιτική εκπροσώπηση απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον δεν μπορεί να παρήσατε η κυρία Άστον. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να καταστήσω ε, σαφές το εξής. Είπα προηγουμένως ότι ε, είναι σαφές ε, το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό. Αλλά αυτό που είπε κάποιος από εσάς προηγουμένως ότι είναι σωστό το ότι στη συνθήκη να υπάρχει μόνο η απαλλαγή για την Κομισιόν και για τους άλλους θεσμούς μόνο η πρακτική. Κοιτάξτε, η πρακτική δεν αντικαθιστά το πρωτογενές δίκαιο και ούτε καν το δίκαιο. Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει ε, κάποια νομική κάλυψη και όχι πρακτική εφαρμογή. Γιατί η πρακτική εφαρμογή μπορεί να αλλάξει και μάλιστα μονόπλευρα. Εγώ λοιπόν θέλω να υπάρχει δίκαιο ε, και όχι ε, πολιτική χάρη, επίδειξη χάρης. Ευχαριστούμε κύριε Μπροκ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση και ιδιαίτερα ενημερωτική για τις εργασίες μας. Βεβαίως ε, δεν ε, τελειώσαμε εδώ, ε, θα συνεχίσουμε, υπάρχει και συνέχεια. Ευχαριστώ όλους τους ερωτώντες, κυρίως τους φιλοξενούμενούς μας. Η επόμενη συνεδρίασή μας, Τετάρτη 14 στις 6 ώρα το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Γεια σας.